Uh, Σας καλωσορίζω στη συνεδρίαση της ε, ε, Επιτροπής Απασχόλησης. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ε, δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεύτερον, διερμηνία. Προβλέπεται διερμηνία σε όλες τις χώρες, εκτός από εστονικά, μαλτέζικα και κροατικά. Τρίτο θέμα στην ημερησία διάταξη. Μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων 10 Οκτωβρίου και 28 Σεπτεμβρίου. Ναι. Και περνάμε στο σημείο 4. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει αρκετό καιρό. Ε, είχαμε σε κάποια θέματα συνεργασία με την ε, Επιτροπή Πολιτισμού. Ο δικός μας, ε, ο στάχτης μας είναι ο κύριος Μπενιφάκη. Του δίνω το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά σήμερα θα σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Ελεγγύης. Πρόκειται για μια νέα πρωτοβουλία. Ο είναι να ενθαρρύνουμε την κάλυψή του από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για τις βασικές αρχές της αλληλεγγύης αλλά και να βοηθήσουμε τους νέους Ευρωπαίους όσον αφορά την απασχόλησή τους, όσον αφορά την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του και να αποκτήσουν και κάποιες σημαντικές εμπειρίες για την καριέρα τους επαγγελματική και όχι μόνο και θα γνωρίζετε ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχουν κάποια πράγματα εδώ που είναι διαφορετικά, ασυνήθιοι. Είχαμε την πρώτη φάση στην οποία είχαμε τις εξαγγελίες του Προέδρου ε, το 2011 την κατάσταση της Ένωσης ε, και στην συνέχεια είχαμε τα οκτώ προγράμματα τα οποία και τώρα τρέχουν. Μετά από την φάση της διαβούλευσης με τους εμπλεκομένους τον Μάιο του 2017 υιοθετήθηκε μια νομική βάση ad hoc και έτσι έχουμε το σχέδιο οδηγίας το οποίο και τώρα συζητούμε η Επιτροπή Πολιτικών Θεμάτων είναι κυρίως ε, αρμοδία επιτροπή αλλά και η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων γνωμοδότησε όσον αφορά κάποια ζητήματα ε, κυρίως θέματα απασχόλησης και κάποιους ε, ορισμούς όσον αφορά ευκαιριακή εργασία και δυνάμει του άρθρου 54 του κανονισμού μας έχουμε εμείς την αποκλειστική αρμοδιότητα. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετική αυτή η πρωτοβουλία. Παρουσιάζονται κάποια πρωτότυπα στοιχεία, δίνεται ιδιαίτερη όθηση όσον αφορά την θελοντική εργασία και κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε απασχόληση η οποία θα βοηθήσει ε, με τυπικές και ε, όχι μόνο μορφές εργασίας στην αλληλεγγύη και ε, επομένως σύμφωνα με διάφορες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών θα έχουμε και συμμετοχή και αυτών. υπάρχουν κάποια προβλήματα θα προσπαθήσω με τροπολογίες να τα διορθώσω. Βλέπετε ότι εδώ βασικός στόχο που θέλω είναι να υπάρξουν εγγυήσεις ότι ε, έτσι δεν θα έχουμε μια κερκόπορτα για κάποιες στρεβλώσεις με το σώμα ελεγγύης. Να δούμε το, να, πώς δεν θα χρησιμοποιούνται οι εθελοντές για άλλους σκοπούς, αλλά θα είναι μόνο ε, για της, ε, για την απασχόληση η οποία έχει καθοριστεί ή θα λαμβάνουν κάποια αμοιβή. Θέλουμε επίσης ε, να μην υπάρχει αντικατάσταση της αμοιβόμενης εργασίας με, την, με τον εθελοντισμό. Άρα θα πρέπει να κωδικοποιηθεί αυτό το πλαίσιο που θα ρυθμίζει τους ε, προσωρινούς εργαζομένους και άρα χρειάζονται κάποιες διατάξεις δεσμευτικές για όσους συμμετάσχουν σε αυτό το σώμα ελεγγύης και θα υπάρχουν και εγγυήσεις ε, ποιότητας. Έχουμε συλλογικές συμβάσεις που θα είναι εφαρμοστές, θα έχουμε άλλες εθνικές διατάξεις όσον αφορά κάποιες θέσεις εργασίας ευάλωτες. Επίσης θα πρέπει να ελευθερούν κάποια μέρτα, μέτρα για τα οποία να καλύπτουν κάποιους δημόσιους οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρχει αμοιβή και θα είναι η εργασία ποιοτική με τις εγγύσεις που προανέφερα. Αυτό θα είναι σημαντικό βήμα πρόοδου σε σχέση με τα όσα σήμερα ισχύουν για τους εθελοντές στην Ευρώπη. και έτσι τώρα θα έχουν και ε, φορείς ε, κερδοσκοπική πρόσβαση στο πρόγραμμα όπως ε, το ζήτησαν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων. Συνοηθήκαμε τους κοιόδες εισηγητές και είπαμε να προχωρήσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα να δούμε τι θα γίνει με τις κοινέ αρμοδιότητες, με την ε, Επιτροπή Πολιτιστικών Θεμάτων. Εκεί υπήρξαν κάποιες διαφωνίες. Θα πρέπει να προωθηθεί και να κλείσει το θέμα, να εγκριθεί το συντομότερο. Όσον αφορά τους εθελοντές, αλλά και την απασχόληση. Ε, θεωρούμε ότι είναι δική μας αρμοδιότητα όλα αυτά. Πάντως, υπήρξε συνεργασία και με τις άλλες επιτροπές Οπότε να καταλήξουμε σε μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση για όταν θα πάμε σε τριμερείς ε, διαλόγους με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Μπενιφέη. Η κυρία Κλούν δεν είναι παρούσα. Θα δω λοιπόν το λόγο στον κύριο ε, που, τον, που την αντικαστά. Ευχαριστώ πολύ. Θα μεταφέρω εγώ την παρέμβαση της συναδέρφου, που δεν μπορεί να είναι εδώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη γνωμοδότησή του, το συντάκτη της δηλαδή. Όντως είναι μια καλή πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και προσφέρει και πολλές ευκαιρίες στους νέους από ολόκληρη την Ευρώπη. Είχε μια καλή εκκίνηση με 3.500 νέους η πρωτοβουλία αυτή, η οποία γράφηκαν και είναι ένα θετικό παράδειγμα υλοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής. Μάλιστα μετά από το σεισμό στην Ιταλία δραστηριοποιήθηκαν πολύ. Υπογραμμίζει επίσης ο ε, συναδελφός ότι θα έπρεπε να υπάρχει ευρωπαϊκή δέσμευση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δηλαδή και να δίνουν την ευκαιρία στους νέους έτσι να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους. Έτσι μαθαίνουν και χρήσιμα πράγματα για την μελλοντική τους ε, σταδιοδρομία ε, αλλά ακόμα κι αν όχι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία γιατί οι νέοι πηγαίνουν σε κοινότητες και υλοποιούν έργα τα οποία είναι θετικά για τις πόλεις, για τις κοινότητες και συγχρόνως ε, κάτι μαθαίνουν το οποίο μπορούν να εφαρμόσουν και σε άλλους τομείς της ζωής τους. Η κυρία Κλούνε λοιπόν εξετάζει τροπολογίες τις οποίες θα υποβάλει αλλά κατά τη γνώμη της η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να ξεκινάει από θελοντική βάση και μαθητεία σε μια αναλογία 80-20 έτσι ώστε το πρόγραμμα να παραμείνει σε θελοντική βάση. Το να περιοριστεί σε μη κερδοσκοπικού σκοπούς ο αθλητισμός μπορεί να είναι κάτι ενδιαφέρον, αλλά έτσι καλώς πρέπει να υπάρχει ε, σχέση με κοινωνικές εταιρείε ε, χωρίς κερδοσκοπικούς σκοπούς. Τέλος, πιστεύει ότι το λεκτικό πλαίσιο είναι κάτι πολύ βασικό για να πετύχει το πρόγραμμα και να μπορέσει να προστατεύσει και τους συμμετέχοντες. Είναι πολύ σημαντικό ένα τέτοιο πλαίσιο να φτιαχτεί, να εκπονηθεί και ευχαριστεί πολύ και τον συντάκτη της γνωμοδότησης και τους σκιώδης εισηγητές και προσβλέπει σε συνεργασία για τη συνέχιση του έργου αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Σιντνάσκα, δεν είναι παρούσα όμως. Υπάρχει κάποιος που την αντικαθιστά. Όχι. κυρία Χάρκιν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να καταφτάσω. Δεν άκουσα την εισήγηση του συντακτή της Έχω διαβάσει όμως τη γνωμοδότηση και πρέπει να πω ότι γενικά Σύμφωνο με πολλές από τις τροπολογίες που έχετε υποβάλει. Νομίζω συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να διαχωρίσουμε τους δύο διαφορετικούς άξονες, να φροντίσουμε να υπάρχει σημαντική διάκριση ανάμεσα, σαφής διάκριση ανάμεσα στον εθελοντισμό και την απασχόληση. Δεν είμαι καν βέβαιη αν θα πρέπει η συγκεκριμένη πρόταση να περιλαμβάνει πτυχή για την απασχόληση. Δεδομένου ότι δεν είναι ακριβώς ε, το ίδιο με την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού και ότι η ε, ισορροπία είναι 80-20%, ε, εάν έχουμε σαφή διάκριση ανάμεσα στην απασχόληση και τον εθελοντισμό, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τον ε, εισηγητή είναι η διάκριση ανάμεσα σε ιδιωτικούς και δημόσιους ε, οργανισμούς. Θέλει να διαγράψει την δυνατότητα ιδιωτική φορείς να μπορούν να εποφελούνται από πρακτική άσκηση εθελοντών. Θα ήθελα να το συζητήσω αυτό περαιτέρω ε, για διάφορους λόγους. Καταρχάς, οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα πληρώνουν για την πρακτική άσκηση. Πρόκειται για πόρους που δεν θα είχαμε εναλλακτικά και είναι δυνατό, είναι πιθανό κάποιοι από αυτούς που επιδιώκουν μια θέση πρακτικής άσκησης να θέλουν να εργαστούν για ιδιωτικούς οργανισμούς. Δεν έχω καταλήξει σε οριστική θέση στο θέμα αυτό. Είμαι ανοιχτή ε, για συζήτηση. Ίσως όμως θα ήταν χρήσιμο να το συζητήσουμε αυτό και να δούμε εάν θα συμπεριλάβουμε ή θα αποκλείσουμε τη δυνατότητα αυτή και αν τη συμπεριλάβουμε να γίνει αυτό με κάποιον τρόπο ώστε να έχουμε τέτοια νομοθεσία ώστε να μην μπορούν να συγκεντρώσουν κέρδη ιδιωτικέ εταιρείε χρησιμοποιώντα ευρωπαϊκού πόρου ε, και να μην ε, του χρησιμοποιούν για ε, λόγου δική του προβολή και διαφήμιση. Επίσης, συμφωνώ με τον εισηγητή ότι χρειάζεται πιο ισχυρή διατύπωση εκεί που μιλάμε για απασχόληση, για θέσεις απασχόλησης και πρακτικής άσκησης θα πρέπει να αναφέρονται στόχοι που συνδέονται με την εκπαίδευση κλπ. Δεν θα παριθμίσω όλους τους λόγους. Ε, απλά ήθελα να σας επισημάνω τι ακριβώς περιμένουμε εμείς ε, από το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, όσον αφορά την ενιαία δικτυακή πύλη, τίνω να συμφωνήσω με την ιδέα. Νομίζω ότι είναι χρήσιμη ο κόσμος ξέρει τι ψάχνει. Γίνεται πολλή δουλειά στον τομέα αυτών Και θέλουμε να φροντίσουμε να μην ε, βάλουμε κατά μέρο τις εργασίες που ήδη έχουν γίνει, θα πρέπει να φροντίσουμε να προσθέσουμε αξία σε αυτά που ήδη γίνονται στον τομέα αυτών. ένας από τους τομείς όπου μάλλον έχω διαφωνία ή που θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω είναι η τροπολογία 18 όπου αναφέρεστε στην ε, πλήρη ή μερική ε, απασχόληση στον εθελοντισμό ή αναφέρεστε και στον ελεύθερο χρόνο. Ε, θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό περαιτέρω ε, την τροπολογία 19 σας ε, την στηρίζω. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε να, ότι δεν θα υπάρξει υποκατάσταση πληρωμένης εργασίας, ε, αλλά νομίζω ότι οι βοηθοί μας ήδη το συζήτησαν αυτό. Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και προσλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή και με τους σκιώδεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι κατάλαβα, ο κύριο Χέτμαν αντικαθιστά την κυρία Ζητνάνσκα. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, jeśli koleżanki i koledzy pozwolą, e, kilka słów. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Έχω ασχοληθεί και εγώ με το έγγραφο αυτό και πρέπει να σας πω ότι η γνωμοδότηση αυτή είναι αρκετά λογική και ο συγγετής έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Πράγματι. Μπορώ να συμφωνήσω λοιπόν μαζί του. Στηρίζω και εγώ την ιδέα αυτού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που να βασίζεται στον εθελοντισμό. Όπως επίσης και η ιδέα της απασχόλησης μου αρέσει εδώ. Και εξεπλάγει λίγο από την ροπή που έχει πάρει αυτή η συζήτηση, γιατί κάποιοι φαίνεται να θέλουν να εγκαταλείψουν την ιδέα της απασχόλησης, της άσκησης και των ασκούμενων. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα αυτή. Γιατί έτσι διδάσκουμε στους νέους ε, πώς να συμπάσχουν με τους άλλους και πώς να μαθαίνουν και τη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό για την Ήπειρό μας. Οποιαδήποτε λοιπόν ιδέα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, η έννοια για να βοηθήσουμε την νεολαία μας, πρέπει να έχει συγκεκριμένη διάσταση. Κάθε θέση απασχόλησης που δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χρυσάφι. Και πρέπει να ξέρει ο κόσμος αυτός επίσης ότι του σκεφτόμαστε. Ότι μας ενδιαφέρει να αποκτήσουν και νέες δεξιότητες, αλλά μας ε, ενδιαφέρει και πώς θα χρησιμοποιήσουν στην πράξη τις δεξιότητες που ήδη διαθέτουν και τα προσόντα που ήδη διαθέτουν και να ξέρουν ότι έτσι ε, μπορούν να βρουν μια πρώτη δουλειά ίσως. Που είναι πολύ σημαντικό για την Ήπειρό μας. Θέλω λοιπόν να σας ενθαρρύνω να σκεφτείτε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύες σαν έναν τρόπο για να εκφράσει την αλληλεγγύη του κανείς και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην ανεργία στις χώρες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αντες Λόπες, παρακαλώ. Α, συγγνώμη, ναι. Επανέρχεται ο κύριος Έτμαν. Συγγνώμη, πρόεδρε. Δεν αντικαθιστώ κανέναν ευρωβουλευτή από το ECR. Εγώ είμαι από το ΕΛΚ, έτσι και ασχολούμε με την υπόθεση αυτή έτσι κι αλλιώς. Ναι, ωραία. Τώρα κύριο Πιμέντα Λόπες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μετά από αυτή τη μικρή σύγχυση που ξεκαθαρίστηκε τώρα, πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να αναφερθώ σε αυτό το κείμενο περισσότερο και όχι στους γνωμοδότηση του γιατί Η τελευταία παρέμβαση ακριβώς δείχνει τις διαφορές που έχουμε μεταξύ μας και τους φόβους μας. Εξάλλου, χτες, στα πλαίσια ε, πρωτοβουλίας, μιλήσαμε για την αδήλωτη εργασία, για την παράνομη εργασία και για την χρήση της έννοιας του εθελοντισμού που χρησιμοποιείται μερικές φορές για να αντικαταστήσει πραγματικές θέσεις απασχόλησης. Και ακριβώς αυτό είναι που εξηγεί το τι κρύβεται από πίσω, ποιες είναι οι προθέσεις της πρότασης αυτής. Δηλαδή, τελικά, η μη αμοιβόμενη εργασία, η δωρεάν προσφορά εργασίας δίνει την αίσθηση ότι εκφράζουμε την αλληλεγγύη μα. Στην πράξη όμως αυτό είναι λάθος, δεν ισχύει. Έχουμε διαφορές λοιπόν όσον αφορά ε, τα προγράμματα, τι προτάσεις. Διαφωνούμε με την ιδέα που λέει ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε ε, στη βάση της ελεγγύης. Δεν είναι αλήθεια. Γιατί αν σήμερα έχουμε μια τόσο βαθιά κρίση όπως αυτή που έχουμε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή οφείλεται στην έλλειψη αλληλεγγύης όχι μόνο απέναντι στους λαούς και στους ανθρώπους αλλά και μεταξύ χωρών. Επίσης έχουμε και επιφυλάξεις για το πρόγραμμα που μας προτείνεται γιατί δεν φέρνει τίποτα καινούριο. Οι στόχοι του ευρωπαϊκού αυτού σώματος εθελοντισμού βρίσκονται και αλλού. Ο εθελοντισμός στο εράσμος, η Νέη Ενδράση, η Ευρώπη για τους πολίτες και θα μπορούσα εδώ να αναφέρω και ένα σωρό άλλα προγράμματα ε, τα οποία σε ένα μεγάλο βαθμό καλύπτουν τους ε, στόχους και το πλαίσιο του προγράμματος που συζητάμε. Εδώ λοιπόν πρόκειται για καμουφλάρισμα και δεν έχει καμιά σχέση με την αλληλεγγύη που ακούσαμε πριν. Και επιτρέψτε μου να σας πω ακόμα ότι αυτό το σχέδιο μας υπενθυμίζει τη δημιουργία άλλων ευρωπαϊκών σωμάτων νέων που κατά το παρελθόν παρουσιάστηκαν σε μια σχολή ενιαίας σκέψης. <coughs> Όσον αφορά την πρόταση αυτή καθεαυτή, συμφωνούμε με τις ανησυχίες που εκφράζει ο συντάξης της γνωμοδότησης. Πιστεύουμε και εμείς ότι οι τροπολογίες του εισηγητή είναι θετικές και δεδομένων των ε, ορίων που έχουμε εμείς στην Επιτροπή μας απασχόλησης και των περιορισμών απέναντι σε αυτό το έγγραφο, έχουμε ελάχιστα περιθώρια λοιπόν. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγνώμη, της Επιτροπής Πολιτισμού που λέει ότι ο εθελοντισμός θα καταργήσει τελικά ε, την άσκηση, αυτό είναι κάτι καλό που αναφέρεται. Οπότε εμεί είμαστε κατά της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως συμφωνούμε με τις προτάσεις του εισηγητή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος δεν είναι εδώ. Ο κύριε Μαρτάνσης έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εκτίμησα πολύ αυτά που είπε ο κύριος Μπενιφάη για το Ευρωπαϊκό Αυτό Σώμα Αλληλεγγύης και εκτίμησα πολύ και τις ρήτρες ασφαλείας που θέλει να λάβει για να προστατεύσει τους νέους μας αφενός και αφετέρου να αφήσει την πρωτοβουλία στις χώρες μέλη. Είπε βέβαια ότι οι κανόνες για τα εργασιακά, την ε, εκπαίδευση κτλ. Ε, είναι θέμα των χωρών μελών. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Από εκεί και πέρα. Η ανάπτυξη του εθελοντισμού είναι μια καλή ιδέα. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι έχει μια καλή ιδέα η Επιτροπή. Ο κύριος Μπενιφέη όμως νομίζω ότι εξέφρασε και κάποιους φόβους, τα είπε και ο προλαλής σας. <clears throat> και ανοιχτά. Δεν πρόκειται εδώ για νέους 17 με 30. Εγώ νομίζω ότι στα 30 δεν είμαστε πια τόσο νέοι. Μήπως εδώ λοιπόν πρόκειται πραγματικά για ένα μακιγιάρισμα που κάνουμε ένα καμουφλάρισμα για να κρύψουμε τα νούμερα της ανεργίας. Μήπως εδώ θέλουμε να απασχολήσουμε τους νέους μας 17 με 30. Την επόμενη φορά θα βάλουμε τα 35, τα 40. Μήπως δηλαδή τελικά φοβάμαι πρόκειται για κατάχρηση που κάνουμε για να χρησιμοποιήσουμε τον εθελοντισμό ως ένα έργο που προσφέρει κάποιος μη αμοιβόμενο. Μας λένε ότι έτσι όμως αποκτάει εμπειρία κανείς και έτσι μπαίνει στον ε, επαγγελματικό χώρο. Όμως ε, αυτή η άσκηση, η άτυπη θα έχει μετά κάποιο, κάποια επιβεβαίωση, κάποιο χαρτί που να επιβεβαιώνει τι εμπειρίες απέκτησαν οι εθελοντές αυτοί θα μετράει στο βιογραφικό τους. Να λοιπόν ποιοι είναι οι φόβοι μας. Και τελικά, μήπως πρόκειται για μια προσπάθεια επικοινωνίας που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού, για να εξηγήσει ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάτι χρησιμεύει. Αν είναι έτσι, αυτό γίνεται στην πλάτη, στο βάρος των νέων 17 με 30. Αυτή είναι η φόβη μου και ο κύριος Μπενιφόη κατάλληλα έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπορεί να μην τα λέει όπως τα λέω εγώ, αλλά θέλει να βάλει κλίδες ασφαλείας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Σόιντερόβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ επίσης όπως και τον εισηγητή για το έργο του, για τις τροπολογίες του. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ακριβώς για ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για τους νέους, προκειμένου αυτοί να μπορέσουν να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό και να αποκτήσουν έτσι μια επαγγελματική εμπειρία. Είναι δηλαδή μια νέα ευκαιρία, μια νέα δυνατότητα που δίνεται στους νέους ολόκληρης της Ευρώπης να μπορέσουν έτσι να δείξουν την αλληλεγγύη τους, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και να προσφέρουν εθελοντικά έργο. Εμείς εδώ ε, είμαστε για να συζητούμε και για την απασχόληση, για τις ευκαιρίες απασχόλησης. Εδώ κάποιοι είπαν ότι είχαμε ήδη το πρόγραμμα για την εγγύηση για την νεολαία που έχει χρησιμοποιηθεί. Εντάξει, μοιάζουν τα προγράμματα, αλλά αυτό δεν θα ασχολείται κυρίως με τα θέματα της απασχόλησης. Γι' αυτό και συμφωνώ με τις τροπολογίες του κυρίου Μπόνιφάη να περιορίσουμε την θελοντική αυτή εργασία πραγματικά σε έργα εθελοντισμού για να αποκτήσει κανείς εμπειρία, να αποκτήσει κάποια προσόντα και νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος, να κάνουμε δηλαδή διάκριση ανάμεσα στον εθελοντισμό και άλλου είδους εργασία. Στην Επιτροπή Πολιτισμού είμαι σκιώδη εισηγήτρια και θα υποβάλουμε και εκεί οι τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τον εθελοντισμό. Αυτό καθ' αυτό, γιατί εμεί θέλουμε αυτή η υπηρεσία εθελοντισμού δεν θα πρέπει σιγά σιγά να διαλυθεί ή να χάσει τη δύναμή της. Όχι, αντίθετα. Θέλουμε να γίνει καλή δουλειά και τα 20 χρόνια που είχαμε μέχρι τώρα δεν πρέπει να διαλυθούν, πρέπει να συνεχιστούν. Στην πρότασή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια λέει ότι με το νέο αυτό κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης όταν αρχίσει να ισχύει τότε η υπηρεσία θελοντισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελειώνει. Άρα δεν θα συμπεριληφθεί στη νέα αυτή πρωτοβουλία. Δυστυχώς λέω. Γι' αυτό και η Επιτροπή Πολιτισμού θα δουλέψει πάνω σε αυτό και θα παρουσιάσει τροπολογίες για το εθελοντικό σκέλος, το σκέλος ε, εθελοντισμού σε αυτήν την πρόταση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Κύριε Μπενιφάη, για να απαντήσετε στις παρατηρήσεις, στις ερωτήσεις Ευχαριστώ. Όχι, να μην μακρηγορήσω, διότι σας ανέφερα τα βασικά στοιχεία στην πρωτολογία μου και άκουσα αυτά που είχαν να πούν οι συνάδελφοι οι ε, εισηγητές, τους οποίους ε, ευχαριστώ γιατί ήταν πολύ επικοδομητικά τα όσα είπαν στη συζήτηση μια που ε, τόνισαν όλα τα σημαντικά σημεία. Και γενικώ είμαι ικανοποιημένο από τι θετικέ αντιδράσει και οπότε θα δούμε τα σημεία στα οποία υπάρχουν κάποιε διαφορέ, πώ θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια κοινά συμπεράσματα. Απλώ να σα προσθέσω δύο συγκεκριμένα πράγματα. Δύο σημεία που έδειξαν οι συνάδελφοι. Πρώτα πρώτα να διευκρινίσουμε στην κυρία Χάρκιν και να κάτσουμε να συνεργαστούμε επ' αυτού, να της πω ότι δεν είναι θέμα διαχωρισμού ιδιωτικού και δημόσιου ε, τομέα στην εκθεσή μου. Απλώς ε, των ε, φορέων, των νομικών προσώπων που έχουν κερδοσκοπικό και εκείνων που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Γι' αυτό είπαμε ότι θέλουμε να υπάρχει εθελοντισμός και να μην υπάρχει αποκόμιση κέρδους από τη δουλειά των εθελοντών και το θέμα είναι κατά πόσον θα υπάρχει αμοιβή για ένα στάζι, για κάποια εργασία. Είναι περίπλοκο το θέμα. Θα πρέπει να κάτσουμε και να συνεργαστούμε και να καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις, σε κάποιους καλύτερους ε, συμβιβασμούς. Επίσης έχουμε και την τροπολογία υπαριθμών 23. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Μαρτέν ε, και εδώ έχουμε συγκεκριμένη μνήμα για το θέμα της ε, πιστοποίησης και του στόχου της. Αυτό ήταν ένα αίτημα έντονο από τις νεολαίστικες ε, οργανώσεις και είπαμε ότι θα πρέπει κάπως να αναγνωριστούν οι μη τυπικές, οι μη κλασικές δεξιότητες και πάλι να ευχαριστήσω τους σκιώδεις συζητητέ για τα όσα είπανε ε, και για τη δουλειά τους. από κοινού θα γεφυρώσουμε τις διαφορές μας όπου υπάρχουν. Πάντως, αυτές εξ αρχή ε, ε, είπαμε ότι συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή του καλύτερο τρόπο και ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος για να μας σχολιάσει εάν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ο κύριος Όιμπε ή η κυρία Βέλα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέγομαι Φανχάρτε από την Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Θα κάνω κάποιες ε, πρώτες παρατηρήσεις και κατόπιν Ματσούπερ θα αναφερθεί στην πτυχή που άπτεται της απασχόλησης στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις και την ε, γνωμοδότηση αυτή. Πολύ χαιρόμαστε που έχουμε μαζί σας αυτή τη συζήτηση και που έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις παρατηρήσεις σας. Και είμαστε ευγνώμονες που έχουμε σύντομα τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις. Προτού περάσω στα βασικά, θα ήθελα να ε, σχολιάσω δύο παρατηρήσεις όπου νομίζω ότι απαιτείται διευκρίνηση. Καταρχάς, όσον αφορά ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θελοντισμού, εκτιμούμε πολύ τις εργασίες της. Και οι ευρωβουλευτές είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά που γίνεται. Και είναι αλήθεια ότι μπορεί να μην χρησιμοποιούμε πια το όνομα αυτό ως σήμα κατά τεθέν, αλλά έχουμε 20 χρόνια θετικών εμπειριών από την υπηρεσία αυτή. Ε, θέλουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες που έχουμε ε, συγκεντρώσει και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Όσον αφορά την πιστοποίηση και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και στο άρθρο 4 αναφέρεται ρητά ότι περιμένουμε πιστοποίηση της ε, δουλειάς που γίνεται, της εμπειρίας που αποκτάτε. Ε, φυσικά αυτό δεν είναι τυπικό, αλλά δεν πρόκειται για τυπική εκπαίδευση, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει επαρκής αξιολόγηση και επιστοποίηση και της ε, άτυπης μάθησης. Αυτό θα βοηθήσει και τα κράτη-μέλη να αυξήσουν την αναγνώριση όσον αφορά τις εμπειρίες ε, του Σώματος Ελεγγύης. Κάποιες παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν με τη συζήτηση που είχαμε και που αντικατοπτρίζονται και στη γνωμοδότηση του κυρίου Μπενιφέη. Καταρχάς, Έχουμε το θέμα της διασυνοριακής και εγχώριας εθελοντικής δραστηριότητας ε, στο, στην τροπολογία 14. αναφέρεστε στις δραστηριότητες που έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και Εθνική διάσταση. Και επίσης ε, ζητάτε να λαμβάνονται υπόψη και τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, ε, για παράδειγμα, ε, από μειονεκτικά περιβάλλοντα. Δεν θέλουμε να δώσουμε τη σφραγίδα αυτή. Ε, καταρχάς, πέρα από την διεθνική διάσταση, ε, υπάρχει ενδιαφέρον και για τις εγχώριες εμπειρίες και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα από μειονεκτικό περιβάλλον. Δεν θα θέλαμε να αποκλείσουμε ε, νέους που να ενδιαφέρονται, που από την άλλη όμως ε, έχουν την ευθύνη να φροντίσουν άλλα μέλη της οικογένειας τους, ε, ηλικιωμένους κλπ. Επίσης, συχνά άνθρωποι από μειονεκτικό περιβάλλον μπορεί να μην θέλουν να λάβουν τη σφραγίδα αυτή. Θα θέλαμε λοιπόν να μείνει πιο ανοιχτό αυτό και το τελευταίο μας επιχείρημα είναι ότι δεν υπάρχουν εθνικά προγράμματα σε όλα τα κράτη-μέλη και θα είναι χρήσιμο να αποκλείσουμε νέους ή να δημιουργήσουμε ανισότητες ως προς τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους νέους ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους. Ε, θα προτείναμε λοιπόν να συμπεριλάβουμε εδώ και τις ε, εγχώριες ε, τοποθετήσεις. Και Όσον αφορά το ποιοι οργανισμοί είναι επιλέξιμοι, εσείς προτείνατε στη γνωμοδότησή σας, κύριε Μπενιφέη, να γίνεται η διάκριση ανάμεσα σε κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι μη κερδοσκοπικοί μπορούν ε, να έχουν και των δύο ειδών δραστηριότητες ε, και απασχόλησης ε, και εθελοντισμού, όχι όμως οι κερδοσκοπικοί. Εμείς συμφωνούμε με την Γενική Αρχή ότι ε, η ότι ο θελοντισμός δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε υποκατάσταση θέσεων εργασίας. Αυτό φυσικά θα πρέπει να διαφυλαχθεί. Ωστόσο, όσον αφορά τα εχέγγυα, η δική μας θέση είναι ότι η υποκατάσταση θέσεων απασχόλησης δεν εξαρτάται από το είδος οργανισμού, εξαρτάται από τη φύση της δουλειάς που κάνει κανείς. Και προφανώς βλέπουμε να υπάρχει ο κίνδυνος, ε, διότι δεν θέλουμε να προωθήσουμε την μη πληρωμένη εργασία. Αλλά αυτό δεν θέλουμε να γίνεται ούτε και σε μη κυβερνητικού οργανισμούς. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε άλλους τρόπους ε, να μετρούμε την ποιότητα και να γίνεται η πιστοποίηση και να εξετάζονται οι αιτήσει ε, για επιχορήγηση. Δεύτερον, ο στόχος αλληλεγγύης δεν ε, εξαρτάται απαραίτητα από την νομική μορφή ε, ενός οργανισμού. Στο γενικό τοπίο, ενώ στο παρελθόν ήταν πολύ πιο σαφή τα πράγματα, ε, σήμερα βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη ποικιλομορφία, βλέπουμε πολλούς μεγάλους οργανισμούς και ιδρύματα. Από την άλλη, βλέπουμε ε, πολύ μικρούς φορείς ε, να ε, δημιουργούν κοινωνικές επιχειρήσεις για να λάβουν επιχορηγήσεις. ή έχουν άλλες δραστηριότητες για να αντισταθμίσουν κάποιους δημόσιους πόρους που δεν τους είναι πια διαθέσιμοι. Ε, δεν πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, αποκλείσουμε διάφορες δυνατότητες ε, και ναι θα κλείσω. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε μικρούς εθελοντικούς οργανισμούς που εργάζονται στο πλαίσιο μιας ομοσπονδίας. Και ναι, θα κλείσω. Έχουμε ένα σύστημα που επιτρέπει ε, σε επιχειρήσεις ε, να ε, συμμετέχουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επιχειρηματικής ευθύνης. Ζητώ συγγνώμη που χρειάστηκα τόσο χρόνο και ο Μάτς έχει να προσθέσει κάποια πράγματα. Πολύ σύντομο θα είμαι. Από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την γνωμοδότηση αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική στο πλαίσιο της οργανικής ε, διαδικασίας. Ε, φυσικά ε, ακούσαμε ενδιαφέρον αυτά που είπατε για την διάσταση της απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Θέλουμε να επιτρέψουμε στους νέους Θέλουμε να προσφέρουμε στους νέους σε μια νέα σειρά ευκαιριών σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και θέλουμε να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα σε αυτό που κάνουμε. Δεν θέλουμε φτηνό εργατικό δυναμικό και υποκατάσταση θέσεων εργασίας. Επιμένουμε και η πρακτική άσκηση να πληρώνεται ενώ στο Συμβούλιο ήταν ε, μερικοί που επέμεναν να μην έχουμε ε, ε, αμοιβούμενη πρακτική άσκηση. Όλοι είμαστε υπέρ της σαφούς διάκρισης ανάμεσα στις διάφορες δραστηριότητες. Και η τελευταία μου παρατήρηση έχει να κάνει με το χρονοδιάγραμμα. Γνωρίζετε ότι αυτή η πρωτοβουλία ήταν μέρος της κοινή ε, διακήρυξης. Ε, επρόκειτο στόχο είχε λοιπόν να ολοκληρωθεί εντός του έτους. Ε, θα ακούσατε ότι χθε το Συμβούλιο σημείωσε κάποια πρόοδο. Το συμβαστικό κείμενο της Προεδρίας θα πάει στο Συμβούλιο σε δύο εβδομάδες. Τα πράγματα λοιπόν ε, κινούνται γρήγορα και ελπίζουμε ότι και στο, και στο Κοινοβούλιο θα υπάρξει γρήγορη συμφωνία ανάμεσα στις δύο επιτροπές για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε τον εισηγητή που έχει δει στο λόγο. Σε αυτά τα οποία είπατε θέλω να προσθέσω κάτι. Να τονίσω ότι κατά τη γνώμη μου ως εισηγητού για να σας τα πω πάρα πολύ σύντομα. Θα πρέπει αυτά τα προγράμματα να αποτελούν οδηγό για το μέλλον. Αυτό το πνεύμα πρέπει να έχουν όσον αφορά τον εθελοντισμό, όσον αφορά αυτή την περιχαρακωμένη αυστηρά εργασία. Έτσι, να φτιαχτούν τα προγράμματα κατά τη γνώμη μου και θα ήταν καλύτερα, λέω, Εάν έχουμε αυτή την ε, διάκριση με κριτήριο μόνο το κερδοσκοπικό εμεί χαρακτήρα και όχι με άλλα κριτήρια. Τους κι αλλιώς είναι δυνατόν να πληρωθεί αμοιβή και για τους ε, ε, μαθητευόμενους και για τους εργαζόμενους. Τώρα για τα in-country placements ναι, καταλαβαίνω πού το πάτε, αλλά δεν θέλω να υπάρξουν αντικίνητρα στα κρατημέλη που δεν το έχουν αυτό προς το παρόν και άρα να μην το κάνουν στο μέλλον. Γι' αυτό θέλω τα in-country placements να προβλέπονται μόνο για κάποιες κοινωνικές ομάδες μειονεκτούσες. Όποιος το κάνει, το κάνει. Αλλιώς είναι πρόβλημα του κράτους μέλους, είναι δική του ευθύνη. Και ευχαριστώ. Προθεσμία για τροπολογίες 15 Νοεμβρίου το μεσημέρι και πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή μας στις 11 Ιανουαρίου και θα ψηφίσει η Επιτροπή Πολιτισμού στις 23 Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ όλους για όσα είπατε. Πάμε στο σημείο παραδείγμα 5 διατάξεως. Είναι η τροποποίηση του κανονισμού κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σχετικά με το καθορισμό των τυποποιημένων κλιμάκων με δύο κόρπου για, για τα κατοπολιτική ποσά για επιστροφή δαπανών κρατών μελών από την Επιτροπή προ τα κράτη-μέλη. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Στον κύριο Ντι Πιετραντώνιο, που είναι ο αρμόδιος τμήματάρχης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τα μέλη και τους βουλευτές για την ανταλλαγή απόψεων. Το θέμα είναι τεχνικό αλλά πολύ σημαντικό για το θέμα το πώς θα πλουστεύσουμε το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δουλεύει στην πράξη και Έχουμε να κάνουμε με την εφαρμογή του άρθρου 14 παραγράφο 1 του σχετικού κανονισμού. Πρόκειται για ένα άρθρο σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μπορεί να προβαίνει σε κατεξοδότηση πράξη, ώστε να ε, εκπληρώνει αυτές τις ενέργειες. Έτσι, δεν υπάρχει ε, πολύ γραφειοκρατία για τα κράτη-μέλη, τι αρχέ. Δεν υποχρεούνται πλέον να αναφέρουν σχετικά με, ε, με αυτές τις δαπάνες, να υποβάλουν ε, τιμολόγια, αποδείξεις, αλλά υπάρχει τώρα συμφωνία ε, για αυτό το μοναδιαίο κόστος βάσει της κλίμακας αυτής και όλα αυτά θεσπίζονται από την κατεξοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε φτάσει τώρα στην τέταρτη τροποποίηση αυτής της νομοθεσίας. Μέχρι τώρα ήταν επιτυχημένη αυτή η ρύθμιση και χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας στήριξε ε, σε αυτή τη ε, διαδρομή τα πρόσφατα χρόνια. Αυτή η κατεξόδηση πράξη επίσης μπορεί να καλύψει κάθε πράξη που ενδιαφέρουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με τις ε, σχετικές αυτές δαπάνες. Και έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις και έτσι έχουμε ασφάλεια δικαίου με την κατεξόδηση πράξη. Γιατί τα κράτη-μέλη μπορούν να είναι σίγουρα ότι θα χρησιμοποιήσουν την επιλογή για την κάλυψη των δαπανών. Επίσης ε, καλύπτονται ε, πρακτικές ε, οικονομικού ελέγχου και λογιστικής. Αυτά από την εξουσιακή πράξη, οπότε και περιορίζεται το deal μεταξύ κομισιών και κράτους μέλους. Και το κράτος μέλος ασχολείται και αναφέρει σχετικά με τους δικαιούχους κάθε φορά και στις δημόσιες προμήθειες και διαγωνισμούς. Ξεκίνησε αυτή η διαδρομή το 2015. Είχαμε την ε, κατευθυντική πράξη η 2195 η οποία δημοσιεύθηκε στις 9 Εβδόμου του 2015 και απλό είναι αυτό το νομικό εργαλείο γιατί προβλέπεται το σώμα της, ε, του που δεν έχει, δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται αναπερίπτωση περίπτωση και αυτό το οποίο αλλάζει σε κάθε τροποποίηση του νομοθετήματο είναι τα παραρτήματα που έχουν τεχνικό χαρακτήρα. Το 2015 στην πρώτη εκδοχή του νομοθετήματο, είχαμε δύο παραρτήματα για τις δύο πρωτοπόρε χώρες που ήταν η Γαλλία και η Σουηδία και εκεί είχαν προταθεί κάποιες ε, απλουστευμένε διαδικασίε για τις πράξει τι οποίε θέλουν να προβούν και έχουμε την πρώτη τροποποίηση του νομοθετήματος το 2016. Οπότε και θεσπίσαμε πέντε ε, μοναδία τέτοια κόστη για Τσεχία και Βέλγιο. Στη συνέχεια ακολούθησε και άλλη τροποποίηση το 2016 με ημερομηνία θέσπιση 31 Δεκάτου ε, για επιπλέον δαπάνες ε, για την Τσεχία και για πρώτη φορά για Μάλτα, Ιταλία, Σλοβακία, Γερμανία και κάτω χώρες. Οπότε φτάνουμε στην τρίτη τροποποίηση της ρύθμισης που τέθηκε, θα τεθεί σε ισχύ με την επόμενη εβδομάδα στις 15 του μηνό συγκεκριμένα. Τότε θα ε, επισημοποιηθεί και 20 μέρες μετά θα τεθεί επισήμως σε ισχύ. Και αφορά τα κάποια κρατημέλη που θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις επιλογές κάλυψης του κόστους. Έχουμε επίσης και κάποιες και νέες χώρες, Ρουμανία, Λιθουανία και κάποιες άλλες, Μάλτα, Τσεχία, Ιταλία και Σλοβακία επίσης για απλουστευμένη κάλυψη αυτών των δαπανών. Επίσης, στην τρίτη αυτή τροποποίηση έχουμε και άλλη μια επιλογή απλουστευμένη για την ε, Σουηδία και τροποποίηση για κάποιους ε, πράξεις προτεραιότητας που αφορούν πρόγραμμα της Σουηδίας. Τέταρτη τροπολογία, τροποποίηση μάλλον, α, συγγνώμη, ε, δεν βγήκε στη διαφάνεια. Αυτό το οποίο σήμερα συζητούμε είναι η τέταρτη τροποποίηση του νομοθετήματο. Θα πρέπει πάνω σε αυτό να ανταλλάξουμε απόψεις και αφορά ε, δύο ρυθμίσει για Γαλλία-Σουηδία, για Γερμανία και για πρώτη φορά για την Κύπρο. Άρα με την τέταρτη τροποποίηση μαζί με την Κύπρο φτάνουμε στις 14 χώρες που χρησιμοποιούν αυτήν την λύση της καταποκοπής κάλυψη του ποσού. Συγγνώμη, υπάρχει ένα πρόβλημα με τα slides. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την οθόνη όπως θα έπρεπε. Τέλος πάντων θέλουμε να συμπλώσουμε τώρα την προηγούμενη τροποποίηση όσον αφορά τη Σουηδία, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παραλείψει ε, κάποιο τμήμα της ρύθμισης όσον αφορά κάποιους άξονες προτεραιότητες για το λειτουργικό πρόβλημα για την Σουηδία και επίσης ε, έχουμε την πρωτοβουλία απασχόληση των νέων που θα αφορά τη Γαλλία και εκεί υπήρχε κάποιο αναπρόσωπο ε, κάποια αύξηση του μοναδιαίου κόστους της αποζημίας από 3.600 στα 4.600 περίπου και είπαμε ότι έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα την πρωτοβουλία απασχόληση των νέων. Στην τέταρτη τροποποίηση έχουμε τρεις νέες ρυθμίσεις για κάποια σχολεία ε, στην ε, Γερμανία που θα αφορούσαν την κοινωνική ένταξη. Θα καλυφθούν τώρα με αυτές τις επιλογές κάλυψης των δαπανών και δύο μέτρα για την Κύπρο πάλι όσον αφορά ένταξη και εκεί ρυθμίζονται κάποιο είδους ημερήσεις και οριές αποζημιώσεις για τα σχετικά μέτρα και άλλη μια ρύθμιση για την λειτουργία της ε, κεντρικής ε, διοίκησης ε, κοινωνικής προνοίας και έχουμε εδώ πέρα κάποιο είδους κλίμακες που συνδέονται με τον μισθό Τεχνικά φαίνονται αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, πάντως ε, υπάρχει μεγάλη διευκόλυνση για τις αρχέ των κρατών μελών μέσω της ε, απλούστευσης. 14 είναι οι χώρε που καλύπτουμε τώρα και πάμε στα 7 δι που θα εκταμιεύσει το κοινωνικό ταμείο με αυτή την πολιτική. Και δεν μιλούμε για πείραμα τώρα πια έχει γίνει πραγματικότητα η απλούστευση στην πράξη και γι' αυτό και θέλουμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα και για την περίοδο 14 έως 20 και έτσι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά και για την επόμενη περίοδο μετά το 20 και για το επόμενο πολιετές ε, πλαίσιο έχει βοηθήσει για τον κανονισμό μου στο Κοινοβούλιο, γιατί έτσι τώρα έχουμε περισσότερες ε, ε, δυνατότητες και πέραν του Κοινωνικού Ταμείου, στον κανονισμό των κοινών ε, διατάξεων και πάλι να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προηγούμενε τροποποίησεις, αλλά και για την συζητούμενη, την πιο τελευταία. Ε, ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρο. Ο κ. Πυρίνσκι έχει δει στο λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή. Και πιστεύω ότι είναι καλό που βάλαμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη, ακριβώ για τους λόγους που τονίσατε κι εσείς. Ότι η πρακτική απλοποίηση είναι πολύ σημαντική για τους δικαιούχους. Υπάρχει ενδιαφέρον και μέσω της δικής μας Επιτροπής θα έπρεπε να στηρίξουμε την παρετέρω εφαρμογή. Θα ήθελα να ζητήσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής το εξή. Πιστεύει πως θα ήταν καλό να πάμε περισσότερο μακριά από αυτό που κάνουμε σήμερα και στον κανονισμό Omnibus που καλύπτει επίσης το άρθρο 14 του κανονισμού αν δεν κάνω λάθος, συζητήθηκε να συμπεριληφθεί ένα κείμενο το οποίο θα αποτελεί σημείο αναφοράς και θα βοηθάει τους δικαιούχους εν δυνάμει να μπορέσουν να βρουν το δρόμο τους για το πώς θα μπορέσουν να εφαρμόσουν την απλοποιημένη διαδικασία. Θα μπορούσατε να προσθέσετε κάτι γι' αυτό ώστε να είναι ενημερωμένη η Επιτροπή μας. Σίγουρα υπάρχει συνδυτοποίηση ότι θα υπάρξει αλλαγή στο συγκεκριμένο άρθρο. Να δώσουμε το λόγο. Ποιος θέλει το λόγο άλλος. Α, ναι, κύριε Χάρκιν. Και μετά να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Η κύριε Χάρκιν. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του ο οποίος μου ζήτησε να σας πω ότι θα έχει τεχνικές τροπολογίες, σας ευχαριστεί. Δεν ε, βλέπουμε κανένα πρόβλημα. Χαιρόμαστε για τον κατάλογο των χωρών, αλλά έχει την εξής ερώτηση. Τι είδους στοιχεία στέλνουν οι χώρες μέλη ώστε να γίνεται ο υπολογισμό του τυποποιημένου του μοναδιαίου κόστους. Και εσείς περιοδικά αυτόματα κάνετε την αναθεώρηση και ένα προσωπικό σχόλιο. Βλέπω ότι το 50% των χωρών χρησιμοποιούν τις απλοποιημένες διαδικασίες. Γιατί Έχουμε πει ότι υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και ρωτάω την Επιτροπή υπάρχει πιθανότητα και άλλες χώρες μέλη υπάρχει κάποιο τέτοιο σήμα που να στέλνουν ότι θα περάσουν και αυτές σε αυτή την απλοποίηση. Ωραία, για να προσπαθήσετε να απαντήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις και τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Πρώτον, να απαντήσω στον κύριο Πυρίσκη. Έχουμε το τελευταίο τριμερή διάλογο με την Επιτροπή Απασχόλησης, τουλάχιστον και το Συμβούλιο, και έτσι αποτελεί μέρος της νομοθεσίας που προτείνεται πια. Οπότε έχουμε συμφωνήσει στον τριμερή διάλογο και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί οι τριμερείς διάλογοι στόχο έχουν όχι μόνο να συμφωνηθούν τα απλοποιημένα μέτρα, αλλά να επεκταθούν επίσης και σε όλα τα διαθροτικά και επενδυτικά ταμεία, ώστε όλα αυτά τα ταμεία να έχουν απλοποιημένες διαδικασίες. Οπότε το επιβεβαιώνω και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι όντως ε, γίνονται θετικές ε, παρατηρήσεις όσον αφορά την ε, επιτυχία των ε, συζητήσεων του τριμερούς διαλόγου. Τώρα για την ερώτηση της κυρίας Χάρκιν <clears throat> για τα δεδομένα. Οι χώρες μέλη μας δίνουν ιστορικά δεδομένα. Δηλαδή δεν είμαστε εντελώς αυθαίρετοι. Υπάρχουν κάποια κόστη τα οποία βασίζονται στα ιστορικά δεδομένα ελέγχου που έχουμε από τις χώρες ε, μέλη και ελεγκτές συμμετέχουν στη διαδικασία. Οπότε πριν καταλήξουμε σε κατεξουσιοδότηση πράξη έχουμε τη διαβεβαίωση ότι τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται σε πραγματικό κόστος και μπορούν να το υποκαταστήσουν. Αυτή είναι η βασική απλοποίηση. Αυτή είναι λοιπόν μία προσέγγιση. Επίσης πρέπει να αφαιρθώ και σε μια άλλη προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στην τρίτη τροποποίηση ε, της ε, κατεξουδότησης πράξης και είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια απλοποιημένη διαδικασία για δαπάνες στην εκπαίδευση. Είναι διαφορετική εδώ η προσέγγιση γιατί έχει να κάνει με τα δεδομένα της Eurostat όσον αφορά ε, τους συμμετέχοντες σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης ίσκετ επίπεδα, όπως τα λέμε, και τα, τα διάφορα κόστη που δίνουν οι χώρες μέλη είναι ένα επίπεδο και τα χρησιμοποιεί Eurostat. Οπότε έτσι έχουμε φτιάξει αναχώρα πίνακες με την αναλογία κόστους που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε χώρα, μπορεί, δεν είναι υποχρεωμένη, σε θελοντική βάση για να ακολουθήσει αυτή την απλοποίηση. Ναι, όντω. πρόκειται για τις 50 χώρες μέλη, 50% των χωρών μελών. Ε, ήδη υπάρχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον και θεωρούν ότι είναι επιτυχία χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτή την απλοποιημένη διαδικασία. Τώρα για τις υπόλοιπες χώρες που δεν συμμετέχουν ε, προς το παρόν αλλά δείχνουν ενδιαφέρον φροντίζουμε εμείς και πηγαίνουμε, τους εκπαιδεύουμε, τους ενημερώνουμε, τους εξηγούμε, τους δίνουμε στήριξη χάρη στους συναδέρφους εδώ να έχετε εδώ δεξιά μου έναν από αυτούς ώστε να πάρουν τελικά την απόφαση να ακολουθήσουν και αυτές την απλοποιημένη διαδικασία. Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι στο μέλλον θα συμμετέχουν όλο και περισσότεροι. 35 100 του ESF πιστεύουμε το 2025 θα εμπίπτει σε αυτή την απροποιημένη διαδικασία. Κάτι το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας εν μάλιστα των νέων δημοσιονομικών προπτικών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. Η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων 13 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Απασχόλησης και η προθεσμία για αντιρρήσεις από πλευράς του Συμβουλίου ή για αίτηση για παράταση της προθεσμίας είναι 20 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Χθες ε, έγινε μια πολύ ζωντανή και ενδιαφέρουσα συνάντηση, ένα γεύμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα αυτή η εκδήλωση. Σήμερα θα συζητήσουμε το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή μας. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Ο κύριος Περέλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι παρόν, όμως, ο κύριος Κυρέλ. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Ιβ Καλτέ, που είναι ο Γάλλος αντιπρόσωπος και συμπρόεδρος της πλατφόρμας. Παρακαλώ, κύριε Καλτές, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω θα έρθει ο κύριος ε, Κουρέλ γιατί από κοινού θα κάναμε αυτή την ε, παρουσίαση γιατί έχουμε τα θέματα τα δημοσιονομικά και τα λειτουργικά της πλατφόρμας και είπαμε εγώ να σας κάνω έναν πρώτο απολογισμό από πλευρά της υπηρεσίας μας και από πλευράς Γαλλίας δύο φορές να μιλήσω πρώτα πρώτα να σας πω ακριβώς ε, ποια υπηρεσία εκπροσωπώ να σας ε, κάνω έναν απολογισμό για την πλατφόρμα και για τα προβλήματα, τις προκλήσεις που έχουμε ακόμα. πρόσωπο λοιπόν ε, της ε, Γαλλίας και συμπρόεδρος επί πέντε έτη για αυτή την απασχόληση που είχε και κάποιο θελοντικό χαρακτήρα, φιλανθρωπικό και Μερική απασχόληση για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την μεταρρύθμιση για την επιθεώρηση εργασία στην ε, Γαλλία και να μπορέσουμε πιο αποτελεσματικά να ε, καταπολέμησουμε την παράνομη εργασία με ειδικέ ε, διοκτικέ ε, ομάδες και έτσι να είμαστε όπω λέγαμε πιο αποτελεσματικοί συνεχίζω να εκπροσωπώ την Γαλλία και συνεχίζω να εργάζομαι στην επιθεώρηση εργασίας. Τώρα, το, η υπηρεσία μας ε, έχει έναν πρόεδρο, δύο αντιπρόεδρους. Ο Λουίς Ρενάρς είναι ο συνάδελφος και προσωπεί την Λετωνία. μετέχει, σε εργασίες ε, του γραφείου μας με τους συνεργάτες του και είμαστε σε στενή συνεργασία. Και θα πρέπει να αναδείξουμε τώρα την ποιότητα της συνεργασίας μας και της συνεργασίας των συμπροέδρων. Δεν είναι διακοσμητικός ο ρόλος μας. Οι προτάσεις μας λαμβάνονται υπόψη για το έργο της πλατφόρμας και έχουμε είτε τηλεσυνεδριάσεις είτε ε, τα λέμε από κοντά και προσαρμόζουμε στις ανάγκες το πρόγραμμα των εργασιών μας. Για να δούμε τώρα τα αποτελέσματα της πλατφόρμας. Υπάρχει μια έρευνα ε, για το αν υπάρχει ικανοποίηση συμμετέσχουν τα τακτικά μέλη και η κοινωνική εταίρεια. Είχαμε το 17-5 ερωτηματολόγια, είχαμε 28 απαντήσεις και προέρχονται από 23 κρατημέλη. Το ερωτηματολόγιο έλεγε αν υπάρχει κάποια πρόοδος όσον αφορά τους τεθέντες ε, στόχους, όσον αφορά την αποστολή της πλατφόρμας, οπότε μετά κάποιους μήνες λειτουργίας οι απαντήσαντες είπαν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και 43% των απαντήσεων είπαν ότι θεωρούν προς τα επιτευθέντα αποτελέσματα είναι καλά ή πολύ καλά. 46% είπαν ότι υπάρχει μέτρια, συγκρατημένη πρόοδος. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ε, εν μέρη διαπίστωση επιτυχίας, εν μέρη ε, διαπίστωση μικρότερης επιτυχίας, τόσο συγκρατημένες... και με την πλατφόρμα αναπτύσσουμε μια προβληματική που ικανοποιεί κυρίως όσον αφορά το ότι έτσι έχουμε ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών για το κάθε κάτω μέλος έχει άλλες μεθόδους. Αυτό θεωρείται πολύ παραγωγικό για όλους μας και έτσι μπορούμε καλύτερα να καταλάβουμε πώς εργάζονται οι συνάδελφοι και επίσης πώς αντιμετωπίζουν τα διάφορα ε, θέματα και παίρνουμε ιδέες. Δεύτερο σημείο που υπήρξε ικανοποίηση. Είναι τότε έτσι, έχουμε περισσότερες ε, δεξιότητες ε, από πλευράς των εμπειρογνωμόνων, έτσι γίνονται καλύτερα δηλαδή και έχουν ε, συνταχθεί και κάποιες μελέτες από την πλατφόρμα και έτσι υπάρχει περισσότερη επίγνωση, περισσότερη γνώση των φαινομένων ανά την Ευρώπη. Τι γίνεται δηλαδή σε κάθε μία από τις χώρες μας. Εκεί που είχαμε πιο συγκρατημένη ικανοποίηση ήταν το θέμα των επιπτώσεων του έργου μας για τις επιδόσεις των διαφόρων αρχών για το κατά πόσον βοηθούμε να βελτιώσουν αυτές τις επιδόσεις οι διάφορες αρχές. Κατανοητό και επίσης για το πόσο έχει μπορέσει η πλατφόρμα να εκπαιδεύσει τα κράτη-μέλη ή τέλος πάντων να κάνει τα κράτη-μέλη να αναβαθμίσουν τις επιδόσεις τους και την πολιτική τους. Θεωρήθηκε ότι είναι χρήσιμη η πλατφόρμα κυρίως γιατί έτσι ε, κατά 93% είπαν ότι υπάρχουν καινούργιες ε, ε, ικανότητες και δεξιότητες από τα μέλη της. Και βελτιώνεται έτσι η διοίκηση, η λειτουργία των υπηρεσιών κλπ. Και αυτό ικανοποίησε. Είπαν επίσης οι συνάδελφοι ότι είναι ενδιαφέρον να ακούει ο ένας τον άλλον για ε, το θεματολόγιο μας. Οπότε και είχαμε και κάποιες συναντήσεις τύπου ολομέλειας, είχαμε κάποιες θεματικές ημερίδες, ε, δηλαδή αναπτύξαμε δικτύωση, ε, ήμασταν μαζί δύο μέρες ε, και δουλέψαμε τα θέματα προτεραιότητας. Τώρα, όσον αφορά την εκπροσώπηση κάθε χώρα μέλος, μπορεί να θεωρηθεί ότι έτσι γίνεται καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών για την πλατφόρμα ε, και προς κάποιον οργανισμό τον, τον οργανισμό, την υπηρεσία των ομολόγων και λιγότερο με τις άλλες υπηρεσίες πάντα για το έργο της πλατφόρμας τώρα αποτελέσματα που έχουν διαπιστωθεί Πρώτα-πρώτα λένε τα κρατημέλη ότι χάρη στην πλατφόρμα υπάρχει επαφή με άλλα κρατημέλη και έτσι έχουμε συνεργασία, ανταλλαγή πρακτικών και έτσι αναπτύσσονται κάποια ελεγκτικά κοινά προγράμματα Κάποιε χώρε επομένω ήδη το έχουν κάνει αυτό και κάποιε άλλε είπαν ότι στο άμεσο μέλλον, του επόμενου μήνε, θα κάνουν το ίδιο. Ε, Επίση, προκύπτει σαφώ ότι έμαθαν τα μέλη μα το πώ εξελίσσεται η μεθοδολογία μας για κάθε χώρα. Ας πούμε για την Γαλλία πήγαμε ε, και ήταν πολύτιμο σε μια συνολική αντιμετώπιση του θεματολογίου των θεμάτων μας. Άρα συνοπτικά κάνοντας μια σύνδεση μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αυτή η ανταλλαγή των πρακτικών, των οργανώσεων ε, αναπτύσσονται σχέσεις μεταξύ κρατών μιλών, μεταξύ των ε, συναρμοδίων ε, υπηρεσιών, με τους ομολόγους τους, για τους σκοπούς μας. Και ε, τώρα για το μέλλον έχουμε ως πρόκληση το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματική συνεργασία, ελέγχους, πώς αυτή η συνεργασία, η διασυνοριακή θα έχει καθημερινό χαρακτήρα. Αυτό είναι τώρα η πρόκλησή μας. Έχουμε το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο κινούμεθα και έχουμε και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Ε, αλλά από εκεί προκύπτουν κάποιοι φραγμοί για ανταλλαγή δεδομένων. Κάναμε και κάποια μελέτη που αφορά ακριβώ τους φραγμούς, τα εμπόδια στο ελεγκτικό μας έργο. Και επίσης υπάρχει έλλειψη ευελιξίας σε σχέση με, τις, με την πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν σας ενημέρωσα ότι έχετε πέντε λεπτά ομιλίας ο καθένας, διότι έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ζορντή Κορέλ που είναι διευθυντής για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και πρόεδρος αυτής της πλατφόρμας. Παρακαλώ σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που άργησα. Ε, το επίπεδο όμως των ελέγχων ασφαλείας ήταν υψηλότερο από ό,τι περίμενα. Ο συνάδελφος ε, είπε τα περισσότερα από όσα πρέπει να υποθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η πλατφόρμα αυτή αποτελεί επιτυχία. Οι συζητήσεις ε, με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ήταν επιτυχής και δεν νομίζω ότι θα φέρει κανείς αντίρρηση. Δεν ήταν πάντα εύκολος ο διάλογος, αλλά ήταν επικοδομητικός και τελικά καταλήξαμε σε ένα εργαλείο λειτουργικό. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στην σύνθεση της πλατφόρμας. Προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε όμως δύο συμπροέδρους από κράτη-μέλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι έτσι ε, δίνουμε κατεύθυνση στις ε, ολομέλειες της πλατφόρμας. Το δεύτερο που θα ήθελα να τονίσω είναι η προέλευση των εκπροσώπων των κρατών μελών ε, που είναι πολύ διαφορετική. Έχουμε κάποιους από τα Τελωνία, έχουμε επιθεωρητές εργασίας κλπ. Και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και την παρουσία των ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και όσον αφορά τους διάφορους τομείς. Και αυτό νομίζω δίνει περισσότερο βάθο στι εργασίε τη πλατφόρμα. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Ε, σύντομη ιστορία των όσων ε, έχουν γίνει. Στην αρχή είχαμε κάποια ε, προβλήματα με παιδικέ ασθένειε, να το πω έτσι. έπρεπε να υιοθετήσουμε τον κανονισμό μα, έπρεπε να εκλέξουμε το Προεδρείο. Αυτό όμως προχώρησε πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω την ε, βούληση και το ε, αίσθημα οικείωσης ε, των περισσότερων, αν όχι όλων των μελών της πλατφόρμας. Θεωρούν ότι αυτό είναι ένα πολύ δυναμικό εργαλείο. Προσφέρει μία παλέτα εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Πολύ σύντομα καταφέραμε να υιοθετήσουμε, διότι έχουμε πολύ ευέλικτες μεθόδους εργασίας. Υιοθετήσαμε λοιπόν αυτό που εγώ θεωρώ, αλλά βέβαια αυτό είναι ανοιχτό προς συζήτηση, ε, φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Και αντί να έχουμε τη συζήτηση κατευθείαν στην Ολομέλεια, ε, συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας όπου συμμετείχαν οι ε, συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα κράτη-μέλη κλπ και εκπονήσαμε έτσι ένα πρώτο σχέδιο το οποίο δεν υιοθετήθηκε αλλά συζητήθηκε από την πλατφόρμα και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι το πρόγραμμα εργασίας λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα όλων των μελών της πλατφόρμας. Χωρίς να θέλω να ε, ε, ζωγραφίσω μια υπερβολικά αισιόδοξη εικόνα, νομίζω ότι γενικά μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τα όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Το πρόγραμμα εργασίας ε, λοιπόν για τα δύο χρόνια ε, προβλέπει τρεις προτεραιότητες, ε, συνεργασία για τις κοινέ δράσεις, για την αμοιβαία μάθηση και την διαβίου μάθηση. Αυτοί οι στόχοι στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Θα ήθελα επίσης να πω ότι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί αλλά όπου νομίζω ότι βλέπουμε να υπάρχει πρόοδος και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα σημαντικά σημεία αναφοράς όσον αφορά τον αντίκτυπο του, της πλατφόρμας είναι οι αλλαγές σε εθνικό επίπεδο. Σε πολλά κράτη-μέλη, αν όχι σε όλα, βλέπουμε ότι η προσέγγιση απέναντι στην ε, αδήλωτη εργασία είναι κατακαιρματισμένη. Ο ΙΒ δεν έχει ε, πάντα πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι Ολλανδοί οι συνάδελφοί του. Ε, αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα και αργά-αργά, αλλά εάν καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο και στον τομέα αυτόν, εάν καταφέρουμε τα κράτη-μέλη να έχουν καλύτερη συνεργασία, καταρχάς σε εθνικό επίπεδο, αλλά μετά και σε διασυνοριακό επίπεδο, εάν καταφέρουμε να έχουν πιο ολιστική αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί, νομίζω ότι θα έχουμε πετύχει ε, κάτι πολύ σημαντικό από πλευρά της πλατφόρμας. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα, αλλά ε, καταλαβαίνω πρώτον άργησα και δεύτερον έχει ε, τελειώσει το πεντάλεπτό μου. Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ, δεν υπάρχει πρόβλημα που αργήσατε. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, που ακούσαμε αυτά που είχαν ε, να μας πει και ο κύριος Καλτές και ο κύριος Κυρέλ. Θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα που μας επισκέφτεται. Ο κύριος Πυρίνσκι έχει προσκαλέσει μια ομάδα επισκεφτών, 30 ε, εκπρόσωποι του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βουλγαρίας, από διάφορα μέρη της Βουλγαρίας, φοιτητές, νομική, διοικητικό προσωπικό και άλλοι. Σας καλωσορίζω λοιπόν εδώ στη συνεδρίασή μας. Ελπίζω να ευχαριστηθείτε την επισκέψη του του Λεχθέντος. Ε, να δώσω το λόγο στην κυρία Λίντς που εκπροσωπεί την ΕΤΥΚ και είναι μέλος ε, της πλατφόρμας για την αδήλωτη εργασία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε ένα σχολείο. ε, όπου είχα την καντίνα. Στις 4 ε, αλλάζαμε τα προϊόντα και γύρω στις 6, 6,5, έπαιρνα τι εισπράξεις και τα βάζα στην τσέπη μου. Ήμουνα 16. Τώρα έχω φτάσει στη δεκαετία μου των 50 και εκπλήσωμαι που διαπιστώνω ότι τέτοιες περιπτώσεις εξακολουθούν να είναι πρόβλημα σε πολλές χώρες. Το θέμα της αδήλωτης εργασίας λοιπόν είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε, είναι κάτι πάνω στο οποίο συμφωνούμε, είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με αυτό. Το θέμα είναι πώς θα μοιραστούμε μεταξύ μας τις επιτυχείς εμπειρίες. Στο Βέλιο έχουμε ένα καλό παράδειγμα με την επιθεώρηση η οποία εντοπίζει τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, ποια είναι η πρώτη επιτυχία της πλατφόρμας. Είναι ακριβώς ότι έχετε δυνατότητα να μοιράζεται ο καθένας με τους υπόλοιπους τις ε, καλές εμπειρίες. Όμως από τις συζητήσεις, αυτό επίσης που έχει βγει, είναι ότι πολλά σχετικά με την αδήλωτη εργασία είναι πολύ περίπλοκα και έχουν να κάνουν, και εξαρτάται δηλαδή αυτή η περιπλοκότητα, ακριβώς από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και, από το... και είναι και αυτό ακριβώς που δυσκολεύει και τους επιθεωρητές να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε και τα περί της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Οι Ευρωπαίοι επιθεωρητές θα πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν ε, με κακό τρόπο το ευρωπαϊκό, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Οι εργοδότες, ε, ας πούμε, λέμε ότι πρέπει να συλλέγουν τα δεδομένα, οπότε οι επιθεωρητές δεν μπορούν να τα ελέγξουν. Τέτοιες πρακτικές πρέπει να αλλάξουν και να γίνουν ε, σωστές ε, συστάσεις. Και σίγουρα θα επανέλθουμε και εδώ σε εσά να σας παρουσιάσουμε τα καλύτερα εργαλεία που θα έχουμε φτιάξει στην πλατφόρμα. Πάντως εσείς πάντα υποστηρίζετε τον κοινωνικό πυλώνα, τα κοινωνικά δικαιώματα. Και είναι κάτι που θα συζητηθεί στο Κέτεμπεργκ και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα δράσης για να υλοποιήσουμε όλα αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί καθορίζονται και νέα δικαιώματα. Και ένας από τους στόχους μας είναι όλες οι χώρες μέλη να έχουν για κάθε 10.000 εργαζόμενους μία επιθόρηση, εργασιακή επιθόρηση. Αυτό είναι ο στόχο λοιπόν που θέλουμε και συμφωνούν τα συνδικάτα, κυβερνήσει κτλ. Να προχωρήσουμε λοιπόν, να δείξουμε ότι όντω αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε και να γίνει και με μια προθεσμία να το έχουμε πετύχει αυτό σε όλε τι χώρε μέλη. Γιατί πάντα κάθε παρανομία ε, δείχνει ότι αυτό που κάνει τον ε, καθένα να παρανομήσει όχι, είτε πρόκειται για δηλητή εργασία, είτε πρόκειται για την φορολογία είτε εξ οτιδήποτε, είναι ο κίνδυνος να τον πιάσουν. Τότε σταματάει την προσπάθεια να παρανομήσει. Το άλλο θέμα που θα συζητηθεί και γι' αυτό θα έρθουμε επίσης να ζητήσουμε τη στήριξή σας είναι, είναι η αναθεώρηση της ε, δήλωσης όσον αφορά τη λογοδοσία των ε, εργοδοτών. Γιατί αν μπορούμε κάπου να αλλάξουμε τα πράγματα γρήγορα, είναι αν σταματήσει αυτή η σύγχυση που έχουμε για την πλατφόρμα που πολλοί λένε μα δεν λειτουργεί καλά, εντάξει τι να το κάνουμε, δεν χρειάζεται. Αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να δείξουμε ότι μπορεί να λειτουργήσει καλά. Από πλευράς ε, των συνδικάτων λοιπόν η αδήλωτη εργασία είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει και η πλατφόρμα αυτή μπορεί να βοηθήσει στην επιτυχία. Ε, ο κύριος Στάμπε τώρα, που και αυτός είναι μέλος της πλατφόρμας, έτσι. Ναι, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκλησή σας. Διαβάσαμε το ενημερωτικό σημείωμα τη συνάντησή σας εδώ και ήταν πολύ καλό γιατί δείχνει ότι έχει επιτευχθεί πολύ πρόοδος <coughs> μέχρι τώρα αλλά συγχρόνως δείχνει ότι παραμένουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και είναι δικό μας καθήκον γιατί είναι μια περίπλοκη δουλειά. Λοιπόν, εγώ εδώ θέλω να σας δείξω που βλέπουμε τις κύριες προκλήσεις. Αναφέρονται και στο δικό σας το σημείωμα, αλλά θα το πω και ό,τι το είπε πριν, ότι υπάρχουν πολλές αρχές οι οποίες εμπλέκονται στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Είναι η εργασιακή επιθεώρηση, είναι επιθεωρήσεις ασφάλειας ε, στην εργασία, φορολογικές αρχές, ε, ασφάλειας, σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και υπάρχουν και οι κοινωνικοί εταίροι, απ' την άλλη. Όλοι αυτοί λοιπόν πρέπει μαζί να καταλήξουν κάπου. Και αυτό καθόλου παρασυμβαίνει. Οπότε το κύριο μας καθήκον είναι να φροντίσει η πλατφόρμα αυτή να είναι σε θέση να συναντήσει όλες αυτές τις προσεγγίσεις. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα είχαμε ένα σεμινάριο στη πλατφόρμα για την συνεργατική οικονομία. Η καταπολέμηση δηλαδή της αδήλωτης εργασίας σε σχέση με την ε, συμμετοχική αυτή οικονομία. Και λέγαμε ότι οι φορολογικές αρχές μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Οι εργασιακές επιθεωρήσεις, οι άλλες αρχές ε, εξαιρούνται. Είναι οι φορολογικές αρχές ο κύριος παράγοντας. Ποιο είναι το μάθημα? Ότι να, ένα παράδειγμα που πρέπει να γίνει συνδυασμός των διάφορων αρχών. Όπως ακούσαμε και πριν, υπάρχει προστασία των δεδομένων και η πρόσβαση των αρχών στα αναγκαία δεδομένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια δυσκολία για πολλές χώρες μέλη. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Η πλατφόρμα λοιπόν πρέπει να λειτουργήσει για να δούμε αν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό και όπως ακούσαμε ήδη, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ε, έχει σαν αποτέλεσμα ε, η πλατφόρμα μας να δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας γι' αυτό και να δούμε τι δεδομένα μπορούμε να μοιραζόμαστε. Και πάλι για να υπογραμμίσω αυτό που λέω. Συγγνώμη, δεν ονομάζεται Ευρωπαϊκή Αρχή εργασίας, αλλά αυτό παραπέμπει στην εργασιακή επιθεώρηση. Και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν πρόκειται μόνο για αυτήν. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό όλες οι εμπλεκόμενες αρχές να κάνουν την προσπάθεια από κοινού. Αυτό είναι βασικό. Και κάτι άλλο, και πάλι λυπάμαι που το λέω εδώ, που είναι παρόντες τόσοι πολιτικοί, είναι πολύ σημαντικό η πολιτική να παραμείνει έξω από την πλατφόρμα. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά όσοι συμμετέχουν στην πλατφόρμα έχουν σαν μοναδικό καθήκον την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Γιατί αλλιώς γίνεται θέμητος ανταγωνισμός Αυτό είναι το θετικό, ότι όλοι το βλέπουμε αυτό, όλοι θέλουμε να πετύχουμε το ίδιο. Είναι περίπλοκο, δεν πρόκειται να γίνεται μια στιγμή στην άλλη, θα πάρει χρόνια, αλλά πιστεύω ότι ο στόχος είναι κοινό και όσο παραμένουμε ε, σε αυτόν τον κοινό στόχο ε, μπορούμε και να προχωρήσουμε. Θα σταματήσω παρόλο που δεν εξάντλησα το χρόνο μου. Πρωτότυπο, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και Φυσικά είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Περίνσκι. Τον άνθρωπο που ξεκίνησε τις εργασίες που κατέληξαν τελικά στη δημιουργία της πλατφόρμας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ εκτιμώ την ευκαιρία που μου δίνετε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι βρισκόμαστε εδώ μαζί με όλους τους κοιόδης εισηγητές και πρόκειται για συλλογική προσπάθεια. Ε, για κατανοητούς λόγους θα συνεχίσω στα βουλγαρικά. Καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, προσκεκλημένους μου από την ε, Βουλγαρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Ε, είχατε δύσκολο ταξίδι νομίζω. Ξεκίνησατε πολύ νωρίς το πρωί. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Τώρα λοιπόν όσον αφορά το θέμα μας. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Δύο λεπτά ομιλίας μου δώσατε, οπότε θα πρέπει να είμαι σύντομος. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η δημιουργία αυτής της πλατφόρμας είναι μια θετική εξέλιξη, διότι αρχικά υπήρχαν αμφιβολίες σχετικά με την ε, χρησιμότητά της. Δεύτερον, η αδήλωτη εργασία είναι όρος πολυσχηδής, είναι όρος πολύπλοκος. Χρειαζόμαστε λοιπόν εμπειρογνωμοσύνη πάνω στο θέμα αυτό. Τρίτον, λάβαμε συνειδητά την απόφαση να χρησιμοποιήσουμε τον όρο tackling, αντιμετώπιση, που περιλαμβάνει την επιβολή κυρώσεων, αλλά και ενθάρρυνση της μετατροπής της αδήλωτης εργασίας σε δηλωμένη. Η Έστερ μας είπε ότι έχει αλλάξει η συμπεριφορά λόγω του φόβου κυρώσεων και νομίζω ότι ναι, ε, είναι θετικό το να ενθαρρύνεται η νόμιμη ε, δουλειά. Ακούσαμε τις ε, γνώμες εμπειρογνωμόνων και βλέπετε ότι εκπροσωπούνται διάφορα συμφέροντα στην πλατφόρμα, συνδικαλιστικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι. Έτσι άλλωστε είχαμε συλλάβει και την πλατφόρμα από την αρχή. Να μην υπάρχει εκμετάλλευση της εργασίας, να μην υπάρχει αθέμητος αντιγωνισμός και ο καθένας να πληρώνει αυτά που πρέπει στις φορολογικές αρχές. Τέλος, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι, η πλατφόρμα εργάζεται εντατικά και μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα είναι να επιφέρει αποτελέσματα στα διάφορα κράτη-μέλη στους διάφορους τομείς. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό λοιπόν μας περιμένει. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, θα ήθελα να προτείνω να μείνουμε σε επαφή με την πλατφόρμα, εσείς ως πρόεδρος ενδεχομένως και σε κάνα χρόνο να δούμε τι θα έχει γίνει στο μεταξύ. Σύμφωνα με την εντολή της, η πλατφόρμα θα πρέπει να καταλήξει σε συμπεράσματα, τα οποία θα πρέπει να μετατραπούν σε αποφάσεις. Και γι' αυτό θα ήθελα να επενέσω αυτήν την ε, ομάδα εργασίας που αναφέρατε. Ε, ο συνάδελφος είπε ότι θα πρέπει να μιλάμε για employment, όχι labor. Για, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ε, είναι σκιώδης συγγήτρη. Σας ευχαριστώ δεν είναι το λόγο. Καλημέρα σε όλους, λέει η κυρία Τόμιτσα. Πέρασε ένας χρόνος. Από τότε που ο κύριος Πυρίνσκι με μεγάλη υπομονή ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις ούτως ώστε να συγκροτηθεί αυτή η πλατφόρμα. Σήμερα θα συζητήσουμε για να δούμε ποιες είναι οι επιδόσεις της πλατφόρμας. Τι πετύχαμε. Είπε ο κ. Πυρίνσκι ότι στην αρχή υπήρχαν πολλές επιφυλάξεις. Όμως έχουμε αποτελέσματα ε, όπως όλοι θέλουμε, δηλαδή έχει καταπολεμηθεί αρκετά η παράνομη εργασία. Αυτό είναι το σημερινό συμπέρασμα. Ότι πέτυχε τους στόχους της η πλατφόρμα. Μόλις ενός ετός είναι η πλατφόρμα. Ε, άρα δεν μπορεί κανείς να περιμένει πάρα πολλά. Όσον αφορά τη δική μας πολιτική ομάδα, σημαντικό είναι να δούμε πώς συγκρίνεται η κατάσταση για την δίδυτη εργασία σήμερα σε σχέση με το παρελθόν και να δούμε και τι θα γίνει στο μέλλον. Έτσι θα προκύψει η διαφορά. Πρόκειται για μέσο πολιτικής. Η πλατφόρμα μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε αποτελέσματα θετικά. Αυτό λοιπόν είναι το κριτήριο και όχι το πόσες φορές ε, έχουν συναντηθεί τα μέλη, το πόσες αρχές, πόσες υπηρεσίες έχουν ε, συγκροτηθεί. Πρώτα-πρώτα να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο. και σε εθνικό επίπεδο με πώς θα γίνει το έλεγχος του πού υπάρχει αθλητική εργασία να συνεργάζονται τα θεσμικά χρόνια μεταξύ του. Σήμερα δεν έχουμε βέβαια τόσο πολύ χρόνο για να τα πούμε εκτενώς. Οπότε και εγώ να βάλω τελεία γιατί νομίζω πάντως ότι τα πήγε καλά η πλατφόρμα και νομίζω ότι σε ένα χρόνο πάλι θα πρέπει να κάτσουμε και να κάνουμε την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Δεν ξέρω τώρα αν ε, μπορούμε να υποβάλουμε ερωτήσεις τους προσκεκλημένους μας, αλλά πάντως εγώ θα ήθελα να τους ζητήσω να ε, μας ε, εξηγήσουν με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα τι υπέτυχε η πλατφόρμα αυτή την χρονιά. Κυρία Μάκιντάρ, για το ECR. Πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά τα οποία έχουμε σήμερα Μπράβο προς την Επιτροπή. Και όπως ξέρετε είμαι πολύ φιδωλή στα μπράβο μου. Και νομίζω ότι με πρόεδρο, με επικεφαλή στον κύριο Πυρίνσκι, προχωρήσαμε για την πλατφόρμα και αποφασισμένοι προχωρήσαμε προς την καταπολέμηση της αδειλώτης εργασίας. Καταπολεμούμε την εκμετάλλευση των εργαζομένων και καταπολεμούμε την υπονόμευση των ε, ε, όσων εργαζομένων είναι ε, σύμφωνοι με τον νόμο και επομένως αυτά έκανε στη διαδρομή της μέχρι τώρα η πλατφόρμα και γνωρίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε συγκεκριμένου στόχους, να είμαστε και φιλόδοξοι και ρεαλιστές. Τέτοια προσέγγιση θα ήθελα να δούμε πώς θα έχουμε την εφαρμογή του νόμου, πώς θα έχουμε ανταλλαγή πρακτικών και γνώσεων. Να μην έχουμε μια τυποποιημένη προσέγγιση Φοβάμαι όμως ότι μια πανευρωπαϊκή επιθεώρηση εργασίας προ τα εκεί τίνει. Ακούσατε τι είπε το 93% που απέντησε τώρα το ομολόγιο ε, σε σχέση με το πού τα πήγαμε καλά και πού λιγότερο καλά. Παρακαλώ, αν μπορούμε να υποβάλουμε ερωτήσει, πέστε μα ε, μήπως σε κάποιε χώρε ε, ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι, ενώ άλλε χώρε θεώρησαν ότι έχουν ωφεληθεί λιγότερο από την πλατφόρμα κλπ. Ε, είμαι Αγγλίδα, είμαι Βρετανίδα και ξέρω ότι όπως γράφουν και αυτά τα πληροφοριακά φυλάδια σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε 1,7% του ΑΕΠ το οποίο σχετίζεται με την αδειλωτή εργασία. Σε κάποιες όμως χώρες ε, είναι πολύ περισσότερο αυτό το ποσοστό πάει στο 13% ή περισσότερο. Άρα σε μερικές χώρες του κόσμου είναι πιο οξυμένο. Άρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα έχουμε κάποιο είδου ε, ε, νομοθεσία για αυτή που έχουμε στη χώρα μας για την ε, σύγχρονη δουλεία. Το πώς θα προσαγόνται στην δικαιοσύνη οι ένοχοι. Οπότε θα πρέπει κάποιο σαν την πλατφόρμα παντού να εξηγεί ποιε είναι οι προσπάθειές μας. Άρα πρόκειται για κάποια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει, ας μην την ε, φρενάρουμε από τώρα, ας καταλάβουμε τι μπορούμε να πετύχουμε και να μην κάνουμε το επόμενο βήμα πριν διαπιστώσουμε ακριβώς τι πετύχαμε μέχρι τώρα. Νομίζω ότι είναι η πλατφόρμα κάτι το πολύτιμο και ότι μπορούμε όλοι στην Ευρώπη να ωφεληθούμε από αυτήν. Ευχαριστώ. Τούμ. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ, τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας. Πρέπει να πω και εγώ στην ομάδα των επισκεπτών ότι μπορείτε να είσαστε ικανοποιημένοι από τον Ευρωβουλευτή σας. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά για αυτό το θέμα. Σε αυτή την μακρά συζήτηση πρέπει να ξέρετε, ή εγώ τουλάχιστον, ότι είναι απελπιστικά τα πράγματα. Και με την επικουρικότητα τελικά είναι δύσκολο να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Αλλά φαίνεται ότι τελικά πάει καλά. Και χθε είχα ένα ολόκληρο κατάλογο με ερωτήσει θέλω να ρωτήσω για τη συνεργασία με τι φορολογικέ αρχέ, για την κοινωνική διάσταση που έχει να κάνει με την εργασιακή φτώχεια για τεχνητά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στις χώρες μέλη εξαιτία του ευρωπαϊκού δικαίου, για τις online πλατφόρμες. Δεν συμβαίνει συχνά. Αυτή τη φορά πήρε όλε τι απαντήσει. Οπότε δεν έχω πια να ρωτήσω τίποτα από τον κατάλογό μου. Κάτι που είναι πολύ θετικό. Έχω όμως κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Είναι μια καλή αρχή. Είναι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα δραστηριοτήτων, διαιτές. Το σύστημα ελέγχου όμως έχει να κάνει με τη γενική ικανοποίηση των χρηστών ε, της πλατφόρμας. Οι εμπειρίες, τα αποτελέσματα και συμφωνώ με την ανατόμηση με την ερώτησή σας που είπε ότι κάθε επιτυχία πρέπει να λέγεται, να ακούγεται. Είναι όμως σημαντικό να έχουμε και μια εξωτερική αξιολόγηση, γιατί τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας είναι τα πιο σημαντικά και ότι λάθη και αποτυχίες μπορούν να εντοπιστούν καλύτερα. Οι βέλτιστες πρακτικές τώρα, δεν ξέρω αν έχετε τέτοιε επαφές, αν όχι ας το σκεφτούμε. Βέλτιστες πρακτικέ και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωσης δεν ξέρω, τι ανατολικέ εταιρικέ σχέσεις, για παράδειγμα, χώρε έχουν. Δεν ξέρω. Αν μπορούν να συμμετέχουν, ξέρω εγώ, σε κάποιο σεμινάριο, σε κάποια δομή, δεν ξέρω πια. Η Νορβηγία, Καναδάς, αν έχουν τις πρακτικές να μας δείξουν, καλό θα ήταν. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω. Η κυρία Κούνεβα δεν είναι παρούσα. Την αντικαθιστά κάποιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν μπορεί δυστυχώς η κυρία Κούρεβα να είναι εδώ σήμερα, αλλά θα σας μεταφέρουμε κάποιες ερωτήσεις της. Πρώτον, ευχαριστούμε πολύ για τη συνάντηση αυτή. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε τα συμπεράσματα. Ε, Σημερίζομαι, δίχως άλλο, τη σημασία που έχει το έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα και αυτή την τελευταία χρονιά για την πλατφόρμα συνεργασία των χωρών, οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν κλπ. Χωρίς αφιβολία, το επαναλαμβάνω, ευχαριστούμε πολύ. Όμως, δυστυχώς δεν φτάνουν αυτά για να διορθωθεί η μάστιγα αυτή της αδήλωτης εργασίας για την κοινωνία ολόκληρη και πιο συγκεκριμένα για τους εργαζόμενους. Η διάγνωση δεν συνοδεύεται από αποτελέσματα. Δεν διαπιστώνουμε να υπάρχει μείωση της αδήλωτης εργασίας. Και μάλιστα, τολμώ να πω ότι σε κάποιες χώρες επειδή εφαρμόζεται αυστηρά η πολιτική λιτότητας, η αδήλωτη εργασία αυξάνεται. Όπως και η ψευδο όπως και η άτυπη μερική απασχόληση που αυξάνει σε πολλές χώρες, στη δικιά μου για παράδειγμα στην Ισπανία. Έτσι υπάρχει εργασία που δεν δηλώνεται επαρκώς. Ε, δηλώνονται λίγες ώρες, ενώ έχει προσφερθεί εργασία περισσότερων όρων. Οπότε οι σφορές είναι μειωμένες, οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν τελικά δικαιώματα. Και επίσης βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται οι επιχειρήσεις που χειροτερεύουν τη συμπεριφορά τους. Όλο και περισσότερες περιπτώσεις έχουμε φόρο αποφυγής και φόρο διαφυγής προκειμένου ε, μάλλον μέσω της μη δήλωσης, ε, της μη πληρωμής εισφορών κτλ. Το είδαμε και πρόσφατα με το θέμα των οδηγών φορτηγών πώς συνεχίζει να γίνεται κατάχρηση από εικονικές εταιρείες. Θα μπορούσα να συνεχίσω και να προσθέσω κι άλλα. Τα ξέρετε πάντως. Η κυρία Λίντς το είπε και συμφωνώ μαζί της ότι αν δεν υπάρξει νομοθεσία, επιπλέον νομοθεσία δηλαδή, πέρα από τόσα κάνει η πλατφόρμα, αν δεν προχωρήσουμε στην εργασιακή εναρμόνιση, αν δεν υπάρξει μια εργασιακή αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν προχωρήσουμε και σε φορολογική εναρμόνιση, κάτι το οποίο έχουμε ζητήσει με εκθέσει μα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο δεν υπάρχει ένα σαφή αγώνα για την καταπολέμηση του φορολογικού ντάμπινγκ. αν δεν κάνουμε απλά πράγματα, αν επικυρώσουμε για παράδειγμα τη Σύμβαση 189 για την ε, απασχόληση στο σπίτι του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένα σχέδια στις χώρες μέλη για την καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας, ε, του χρόνου θα έχουμε μία έκθεση συντονισμού ικανοποιητική, με καλές πρακτικές, αλλά θα εξακολουθούμε να βλέπουμε ότι το πραγματικό αποτέλεσμα όσον αφορά την αδήλωτη εργασία δεν υπάρχει. Δεν θέλω να είμαι άγγελος κακών ε, ειδήσεων, γιατί από ό,τι φαίνεται όλοι είμαστε ευχαριστημένοι με την πλατφόρμα. Τέλος, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να μην ξέρουν αν θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση, οπότε δεν βλέπουν τη χρήση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τι τους βοηθάει να βελτιώσουν τη ζωή τους. Ενώ αυτό θα έπρεπε να είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, βλέπω κανέναν εκπρόσωπο των Πρασίνων. Ούτε του EFTD. Α, παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν σας είδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εμείς από το 2015 άρχισαμε τη συνεργασία μας με τον κύριο Πυρίνσκι ως εισηγητή για την καταπολέμηση της δίδοτης εργασίας και έχουμε τώρα αυτό το σύστημα ανταλλαγής πρακτικών και πληροφοριών και έτσι θα έχουμε αποτελεσματικότητα, θα έχουμε συντονισμό για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο θίγει τους πιο ευάλωτους από τους εργαζόμενους. Και επίσης ε, τώρα ε, περνάμε σε άλλο επίπεδο, πιο φιλόδοξο, γιατί πρέπει να ξεπεράσουμε και κάποιες διαθροτικές δυσκολίες. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορεί να ζυγιστεί, να ε, εκφραστεί ποσοτικά η έκταση του φαινομένου και λέμε ότι πάμε στο 21% αλλά αυτό είναι προσεγγιστικό. Από την άλλη, μετά, από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε το ότι τα δεδομένα συλλέγονται πάρα πολύ δύσκολα και επίση δεν μπορούν όλα τα κρατημέλη να ε, δρουν με την ίδια ένταση συνέχεια. Πολλές φορές έχουμε εθελοντική δουλειά πάνω σε αυτά, αλλά πάντως όσα έχουν γίνει είναι σωστά. Σωστό είναι επίσης να υπάρχει ανταλλαγή στις επιχειρήσεις εργασίας για τους ε, σχετικούς ε, αρμόδιους υπαλλήλους. Οπότε και διασυνοριακά θα πρέπει η Ευρώπη να καταπολεμήσει το φαινόμενο γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων και αυτό βοηθάει. Έχουμε επίσης τις ε, μελέτες που αναφέρθηκαν όσον αφορά και τις ε, εικονικές εταιρείες στην Ευρώπη και έχουμε τώρα τη διαδρομή της ε, του 1,5 έτους οπότε προχωρήσαμε και σε αυτή την σε αυτόν τον απολογισμό του τι έγινε. Ε, νομίζω ότι έπιασαν τόπο τα χρήματα των φορολογουμένων τα οποία αναλώσαμε για αυτή την προσπάθεια. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις ε, κυρώσεις. Ε, έχουμε μια αλλαγή πνεύματος, όλα αυτά θα, θα πρέπει, την νοοτροπία Ο, θα πρέπει να το προωθήσουμε αυτό το νέο πνεύμα στις χώρες μας και ε, η μαύρη εργασία ε, οδηγεί στην παραοικονομία και αυτό καταπολεμούμε και νομίζουμε ότι με τη δράση μας αυτή θα μπορέσουμε να έχουμε ένα τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο κύριος Ντομινίκ Μαρτάν ζητεί τώρα για το ΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, βέβαια, μια τέτοια πλατφόρμα για την αδήλωτη εργασία είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και με το παραπάνω. Χρειάζεται κατεπηγόντως, είναι επιτακτική ανάγκη. Μπράβο κύριε Πυρίνσκι, ειλικρινά σας επενώ, διότι θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι αυτοί οι ευάλωτοι εργαζόμενοι θίγονται και όσον αφορά την κοινωνική πρόνοια, την προστασία της υγείας τους, την σύνταξή τους, ε, αλλά και επιχειρήσεις ε, θίγονται. Και έτσι έχουμε τον ανταγωνισμό. Να μην μακρυγορό. Αλλά τα είπαμε και τον Μάρτιο του 2017 και θυμάμαι ότι η Κομισιόν είχε πει να ε, σχολιάστε τις οδηγίες για την παράνομη μετανάστευση. Πώς πάει αυτή η δουλειά, έχουμε αποτελέσματα, η πλατφόρμα ε, είπαμε ότι θα πρέπει να κάνει για τους απεσπασμένους εργαζομένους μία μελέτη. Επίσης μια άλλη μελέτη για τις εικονικές εταιρείε. Ε, και είχαμε πει τότε το Μάρτιο ότι θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν μέχρι το φθινόπωρο του 2017. Έφτασε το φθινόπωρο. Και είχαν διατεθεί ένα εκατομμύριο ευρώ για τις εργασίες σας, για την αδειλωτή εργασία και επίσης υπήρχαν και κάποια προγράμματα στα οποία επρόκειτο να προβείτε ε, σε κάποια επιλογή. Τι έγινε, προχωρήσατε στην επιλογή. Έμεινα στα δύο λεπτά, Πρόεδρε, όπως λέτε. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Χάτσο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αδήλωτη εργασία είναι κάτι αρνητικό με πολλούς τρόπους, όχι μόνο οικονομικά αλλά και ηθικά. Θα ήθελα να τονίσω τα προβλήματα της ευρωπαϊκής νεολαίας που ε, πλήττεται από ανεργία σε ποσοστό 20% και μιλάμε για κάποια εκατομμύρια ανθρώπων που επηρεάζονται από την κατάσταση αυτή. Οι νέοι θα ήθελαν να έχουν μια νόμιμη δηλωμένη θέση απασχόλησης. Αλλά για πολλούς η αδήλωτη εργασία είναι η μόνη ευκαιρία απασχόλησης. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ακριβώς τη ρίζα του προβλήματος. Και να συντάξουμε νόμους που θα κάνουν αυτήν την ε, πρακτική επώδυνη για τους εργοδότες. Νομίζω ότι πολλοί φοβούνται τις συνθήκες ε, στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Φοβούνται τον σκληρό ανταγωνισμό. Και η ερώτησή μου προς τους εκπροσώπους της πλατφόρμας είναι εάν έχουν ιδέες σχετικά με το πώς μπορούν να προσφέρουν ένα μέλλον στην νεολαία μας που πάντα κινδυνεύει από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για παράδειγμα, ο διτός τρόπος εκπαίδευσης, δηλαδή θεωρία και πρακτική, ε, θα ήταν κάτι πολύ χρήσιμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Άγνες Γιονγκέριους, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ακούστηκαν πολύ έπαινοι για τον Γιώργη και την ε, πλατφόρμα στην αίθουσα και θα ήθελα και εγώ ε, να συμφωνήσω με τους επένους αυτούς. Έχω μία ερώτηση σχετικά με την παρουσίασή σας και κάτι που δεν αναφέρεται πώς προοδεύεται όσον αφορά την εκπόνηση ενός ε, κοινού ορισμού, διότι αν θέλετε να συλλέξετε δεδομένα από όλη την Ευρώπη, θα είναι χρήσιμο εάν υπάρχει κοινός ορισμός για να μπορούμε να μετράμε και την πρόοδο στον τομέα αυτών. Θα με ενδιαφέρε λοιπόν να μάθω αν Το συζητάτε αυτό. Ε, επίσης, εάν πιστεύετε ότι μια κάρτα κοινωνικής ασφάλισης ε, θα βοηθούσε, έχετε προβληματιστεί πάνω στο θέμα αυτό και η δεύτερη μου παρατήρηση είναι πιο συγκεκριμένη και απευθύνεται στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή εργάζεστε πάνω στην αρχή εργασίας. Τι μαθήματα, τι μάθατε μέσα στο πρώτο αυτό έτος που να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ε, στο πλαίσιο της αρχής εργασίας της Labor Authority και προς τα άλλα μέλη της πλατφόρμας. Έχετε από αυτό το πρώτο έτος εμπειρίες που θα μας βοηθήσουν στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ακούστηκαν ερωτήσεις και από την κυρία Γιονγκέριο σχετικά με το τι μάθαμε και τον κοινό ορισμό. Η Τέθηκαν και άλλες ερωτήσεις. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Κιουρέλ για να προσπαθήσει να απαντήσει στο όνομα όλων των ε, μελών σας. Ε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας ε, που οργανώσατε αυτήν την συζήτηση. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη ήταν ε, κρίσιμη στην ε, δημιουργία της πλατφόρμας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Πυρίνσκι για την αποφασιστικότητά του. Ε, κάτι που με έκανε να υποφέρω κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, αλλά νομίζω τελικά ε, καταλήξαμε σε καλό αποτέλεσμα. νομίζω ότι έχουμε καταφέρει πολύ καλά πράγματα και θα παραθέσω εδώ τα λόγια του κυρίου Πυρίνσκι που λέει ότι η αδήλωτη εργασία είναι πολυμορφικό φαινόμενο και απαιτεί και ολιστική προσέγγιση. Δεύτερη παρατήρηση, ιδιαίτερα στην κυρία Τόμς. Πρέπει να μετρούμε την πρόοδο της πλατφόρμας ε, ανάλογα με τη μείωση της αδήλωτης εργασίας ε, στην Ευρώπη. Ναι, αυτό φυσικά το γνωρίζουμε όλοι. Η πλατφόρμα δεν είναι απλά μια πλατφόρμα, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Και δεν μπορεί η πλατφόρμα από μόνη της να τα κάνει όλα. Η Έστερα αναφέρθηκε στις κυρώσεις, αλλά ε, δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε τις πλατφόρμες. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε την πλατφόρμα τμήμα ενός συνόλου. και να απαντήσω συγκεκριμένε ερωτήσει. Η κυρία Τόμ αναφέρθηκε στι ιστορίε επιτυχία, ρώτησε σχετικά με τι ιστορίε επιτυχία. Εγώ θα αναφέρω μία, την ε, αξιολόγηση ομοτήμων ε, που έγινε στην Ρουμανία από μέλη του, της πλατφόρμας. Ο Υπουργός της Ρουμανίας ζήτησε εμπειρογνώμονες από την πλατφόρμα να διεξάγουν μια ει ανάλυση της επιθεώρησης εργασίας της Ρουμανίας και να διαπιστώσουν τι λειτουργεί καλά και τι όχι. Και νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να το συνηθίζουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, μια αρχή, για παράδειγμα, ανοίγει τις πόρτες της τελείως ε, σε εμπειρογνώμονες από άλλες χώρες και με βάση ένα ερωτηματολόγιο εξετάζεται η κατάσταση, χωρίς να κρύβουν τίποτα και δέχονται οι εμπειρογνώμονες να συνομιλήσουν μαζί τους σχετικά με πιθανές βελτιώσεις και νομίζω ότι αυτό αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Αυτό δείχνει ε, τον ρόλο της πλατφόρμας. Ε, δεν ε, βρίσκονται το οι εμπειρογνώμονες μας για να υπερασπιστούν τις χώρες τους, όπως σε άλλες συναντήσεις. Προσπαθούν να προωθήσουν όσο γίνεται την πλατφόρμα. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να το αναφέρω ως παράδειγμα βέλτισης πρακτικής. Επίσης, τέθηκε ερώτηση σχετικά με το αν έχουμε κερδισμένους και χαμένους, αν κάποιος ε, αποκτάει περισσότερα από τους άλλους. Εγώ νομίζω ότι ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει. Βέβαια, ε, η ανταπόκριση της πολιτικής στα διάφορα κρατημέλη διαφέρει. αλλά έχουμε για παράδειγμα τον ε, Ιβ, έχουμε την Έστερ και τον Νίλς ε, που ο καθένας ε, συμβάλλει με τις δικές του γνώσεις και εμπειρίες και έτσι ο καθένας μπορεί να αποκτήσει αυτό που θέλει στην πλατφόρμα. Η κυρία Τούμ δεν νομίζω ότι έθεσε συγκεκριμένη ερώτηση. Προφανώς απαντήσαμε πρωτού τη θέση της ερωτήσης. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις γνώσεις που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα. Επίσης, τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με διάφορες προτάσεις. Ε, μπορείτε να τις δείτε στην ε, ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις για κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, πολύ ευχαριστώ θα απαντήσουμε. Όσον αφορά την νόμιμη μετανάστευση, ε, αυτή ήταν τμήμα της διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λάβαμε διάφορες παρατηρήσεις από την πλατφόρμα και προβλέπεται ένα σεμινάριο στις 30 ε, Νοεμβρίου για το θέμα αυτό. Και όσον αφορά τις ερωτήσεις της κυρίας Γιονγκέριου, όσον αφορά τον κοινό ορισμό, είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε. Του χρόνου θα ε, ξεκινήσει τις εργασίες της σε μια ομάδα εργασίας της πλατφόρμας. Θα πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστικοί σχετικά με το τι μπορούμε να περιμένουμε. Πιθανότατα να καταλήξουμε, πιθανότατα, δεν θέλω να προδικάσω τις εργασίες της ομάδας ε, εργασίας, ε, πιθανότατα λοιπόν να καταλήξουμε σε κοινό ορισμό. Αλλά ο νομικός ορισμός σήμερα ε, ορίζεται σε εθνικό επίπεδο. Και όσον αφορά το τι μάθαμε από το πρώτο έτος ε, λειτουργίας μας, ε, θα σας το πούν αυτό και άλλα μέλη της πλατφόρμας. Στην τελευταία μας συνάντηση συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας που θα συνεδριάσει τον Δεκέμβριο με 22 μέλη που θέλησαν να συμμετάσχουν. η οποία θα υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαίρως, εντός της προθεσμίας ε, του Δεκεμβρίου, ε, μια συνολική εικόνα και ο Ιβ είπε ότι γενικά ήταν ικανοποιημένος με τις εργασίες της πλατφόρμας, ε, μπορεί όμως να βλέπει όμως και κάποιες ελλείψεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Εμείς ευχαριστούμε λέει η Πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι μπορείτε όλοι να λάβετε τον ε, λόγο. Ο κύριος Πυρίνσκι πάντως θα κλείσει την ε, συζήτηση. Και να δώσουμε όμως το λόγο πριν τους κοινωνικούς εταίρους που είναι τόσο σημαντική γνώμη τους όταν ε, έχουμε τέτοιες συζητήσεις. Ε, για την πραγματικότητα τις αποφάσεις που έπρεπε να λάβουμε σχετικώς. Έχετε το λόγο. Η κυρία Λίντς καταλαβαίνω πρόεδρε την απογοήτευση ε, κάποιων βουλευτών ε, όντω είναι πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τους εργαζομένους που έχουν αυτή τη δύσκολη επιλογή είτε να μην έχουν δουλειά ή να πρέπει να δουλέψουν παράνομα ιδίω για τους αυτοπασχολουμένους. Οπότε, να, λέμε ότι πέτυχαμε στο έργο μας ως πλατφόρμα. Ε, το θέμα είναι γιατί τα συνδικάτα αναγνωρίζουν την ε, επιτυχία της ε, πλατφόρμας, μα γιατί πρόκειται για ένα βήμα που μπορούμε να αναδείξουμε τα διάφορα προβλήματα που έχουν κουκολωθεί. Να, ας πούμε τι γίνεται με τους αυτοπασχολούμενους, ε, πιλότους, επιβατηγών ε, αεροπλάνων. Σε όλα τα κράτη-μέλη είπαμε ότι προειδοποιούμε, επισημαίνουμε, κοιτάξτε το καλύτερα. Να, ένα βήμα που μπορούμε να καταθέσουμε τα στοιχεία που έχουμε για τα όσα συμβαίνουν. Βέβαια όμως είναι και μια ευκαιρία πλατφόρμα για κάποια κράτη-μέλη ούτως ώστε να ακουστούν και οι δύο πλευρές. επίσης να ακούσουμε κάποιους πετυχημένους στην Ευρώπη που αντιμετώπισαν το ε, πρόβλημα και έτσι είπαμε να ορίστε μπορούν να βοηθήσουν οι εργοδότες, μπορούν να βοηθήσουν τα συνδικάτα ε, και ακόμα καλύτερα να κάτσουν στο τραπέζι της συζήτηση με εκπροσώπους των κυβερνήσεων. Οπότε έτσι μπορέσαμε να δούμε τι είδους διαδικασίες, τι είδους δομές μπορεί να υπάρχουν και αυτά τα ενθαρρύναμε, αυτά τα διευκολύναμε. Τα είπαμε και χτες στο γεύμα εργασίας για κάποιες κλασικές δυσκολίες, δηλαδή τους δυσνοριακούς εργαζόμενους που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες. Και έχουμε και κάποια προγράμματα ε, κατά τον αλφαβητισμό ε, ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά διάφορους ε, φόρους, διάφορα τέλη κοινωνικής πολιτικής, διάφορα θέματα εργασιακών συμβάσεων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Οι εργοδότες ενδιαφέρονται για αυτά. Θέλαν να τα προωθήσουν. Οι εργαζόμενοι από την άλλη μεριά θεώρησαν ότι είναι πάρα πολύ θετικές αυτές οι προσπάθειες. Έτσι ε, υπάρχει θα υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για άλλους στην Ευρώπη και δεν λέμε για ψευτο αυτοαπασχολούμενους πάντως είναι ξεκάθαρο ότι η πλατφόρμα μας βοηθά να δούμε κάποια προβλήματα τα οποία δεν είχαν αναδειχθεί να δούμε πώς θα αλλάξουμε την κατάσταση και αυτές τις νέες αρχές να δούμε με ποια εργαλεία θα θεραπεύσουμε τα όποια κοινά, τα, πώς θα λύσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Τράμπερ. είμαι πολύ σύντομος. Είναι πολύ σημαντικό η πλατφόρμα να είναι ένα βήμα ανταλλαγής ε, πρακτικών και εμπειριών. Λειτουργεί. Αποδίδει τώρα θα πρέπει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Η διαδικασία όμως δεν ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο, δύο χρόνια. Είναι κάτι το συνεχές και τη συνέχεια ξεπηδάνε καινούργιε μόρφες παράνομης εργασίας. Έχουμε πολύ καλό σύστημα πρόνοιας κοινωνικής στην ε, Δανία, ε, αποδοτικές δημόσιες υπηρεσίες, αλλά είναι συνεχής ο αγώνας μας κατά της ε, πάνω εργασίας. Ξέρω κύριε Πυρίνσκι ότι στη χώρα σα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Είναι συνεχή ο αγώνα, οπότε η πλατφόρμα πολλά χρόνια θα έχει δουλειά να κάνει. Δεν ξέρω, παρεξήσατε αυτά που είπε η κυρία Λίντσε. Βέβαια και η εφαρμογή του νόμου είναι πολύ σημαντική. Αλλά θα πρέπει και το να υπάρχει κάποια διευκόλυνση. Δηλαδή, θα πρέπει πολλές εταιρείε να κάνουν τη μετάβαση από τα αδήλωτα στα δελωμένα, στη δηλωμένη, στην νόμιμη εργασία. Έχουν πολλά. Ε, πάρα πολλοί επιχειρηματίε ε, Βέλγοι και μα ρωτήσαν πώ μπορούμε να κάνουμε τη μετάβαση στην νομιμότητα. Ευχαριστούμε. Και ο κύριο Καλτέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιβεβαιώνω αυτά που είπα και νωρίτερα και μετά από αυτά που άκουσα. Επιβεβαιώνομαι σε αυτή την άποψη ότι δηλαδή είμαστε μέσα σε μια διαδικασία η οποία θα αποφέρει καρπούς μεσοπρόθεσμα. Το θέμα που έχουμε βέβαια είναι ο προβληματισμός για τη νέα αυτή αρχή. Να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες, να εντοπίσουμε ποια είναι τα εμπόδια στην καλή συνεργασία μεταξύ των χωρών και την ανταλλαγή δεδομένων. Θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό για να προχωρήσουμε στο έργο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριο Σπυρίνσκι. Πολλά σχόλια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω, γιατί πιστεύω ότι είναι σαφές πως η πλατφόρμα στο λίγο χρόνο που λειτουργεί έχει πετύχει κάτι πολύτιμο. Και αυτό είναι η διάδραση, η συνεργασία για συζήτηση για διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αδήλωτη εργασία. Τώρα πρέπει να περάσουμε από τη συζήτηση σε συγκεκριμένες κοινέ δράσεις σε επίπεδο χωρών μελών. Και αυτό με ομάδες εργασίας όπως αυτή στη Ρουμανία για την οποία ακούσαμε. Οπότε δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα ήδη ακούσαμε. Είμαστε απέναντι σε μια μεγάλη πρόκληση. Θέλω να ευχαριστήσω πάντως όλους, όπως είπατε και εσείς ε, ήδη, όσοι μίλησαν για το δικό μου έργο και εκείνο των συναδέρφων μου που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και στη δημιουργία της πλατφόρμας αυτής. Αυτό το οποίο δείξαμε εμείς με την συνεργασία ε, φάνηκε όταν φτάσαμε στο επίπεδο δημιουργίας της πλατφόρμας, καταλήξαμε σε μια μορφή που λειτουργεί. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύτιμο επίτευγμα αυτό. Και πάλι λοιπόν ευχαριστώ πολύ όλους τους γιώδες εισηγητές. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό τμήμα, ε, πρόεδρε, που δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. Και αυτοί είναι οι εμπειρογνώμονες οι ειδικοί που εργάζονται στην γραμματεία της πολιτικής ομάδας των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, αλλά νιώθω ότι όταν ε, ακούγεται το όνομα κάποιου νιώθεις κάπως ε, περίεργα, δύσκολα. Γι' αυτό δεν θέλω να πω ονόματα, εν περιπτώσει. Αλλά όμως πιστεύω ότι το έργο τους ήταν πολύτιμο των εμπειρογνωμόνων αυτών. Ευχαριστώ επίσης και όλους εσάς που συμμετείχατε στη σημερινή συζήτηση. Πιστεύω ότι η κοινοβουλευτική μας αυτή η Επιτροπή έχει το καθήκον να αποτελέσει το συνδεκτικό κρίκο ανάμεσα στους νομοθέτες και την πλατφόρμα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για την σημαντική αυτή συζήτηση που είχαμε και θα επανέλθουμε βέβαια. Τώρα έχουμε 3-4 λεπτά στη διάθεσή μας πριν το επόμενο θέμα. Θα περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Τέσσελμπλουμ, ο οποίος θα έρθει σε λίγα λεπτά. να παραμείνετε παρακαλώ, να κάνετε ερωτήσεις στον κύριο Ντάσελμπλουμ. Οπότε διακόπτουμε για 3-4 λεπτά παρακαλώ.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

Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε έτοιμοι για την ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε με τον κύριο Ντάσελμπλουμ. Οπότε, παρακαλώ, καθίστε, συγκεντρωθείτε. Έχετε λίγα λεπτάκια ακόμα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αρχίζουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Ντάσελμπλουμ, στην Επιτροπή μας. Όπως γνωρίζετε, δίχως άλλο, συζητήσαμε πολύ μέχρι τώρα στην Επιτροπή μας για την κατάσταση στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά συζητήσαμε πολύ για την Ελλάδα. Και είχαμε ανταλλαγές απόψεων με ε, Υπουργό Εργασία από την Ελλάδα, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Συμβουλίου της Ευρώπης και την Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων της Ελλάδας. Είχαμε και εκπροσώπους ομάδων ειδικών, θεσμών κλπ. Πολύ χαιρόμαστε λοιπόν που σας έχουμε σήμερα μαζί μας, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας εμπειρίες <clears throat> όσον αφορά τα χρόνια αυτά που αφήνουμε πίσω μας. Υπάρχει μέλλον, υπάρχει μέλλον για το ελληνικό ζήτημα. Και είμαστε πραγματικά έτοιμοι να σας ακούσουμε. Δεν ήμουν εδώ όλα τα μέλη της Επιτροπής μας, όπως βλέπετε. Σίγουρα πολλοί από τους απόντες παρακολουθούν από τους υπολογιστές τους ε, την ε, συνάντηση αυτή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που είστε εδώ. Έχετε το λόγο παρακαλώ για μια εισαγωγή την Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε εδώ σήμερα στην κοινοβουλευτική αυτή Επιτροπή Απασχόλησης. Ο μόνιμος οικονομικός διάλογος ε, με μένα πρόεδρο γίνεται βέβαια στην ΕΚΟΝ. Η Επιτροπή Απασχόλησης όμως καταλαβαίνουμε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το ελληνικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξελίξεις στην εργασιακή αγορά. Στις 27 Απριλίου που μας πέρασε ενημέρωσα την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά το ελληνικό πρόγραμμα. Από τότε έχει επιτευχθεί πρόοδος σε πολλά μέτωπα. Η Ελλάδα και οι εταίροι της κατάφεραν να ολοκληρώσουν ε, την αναθεώρηση του δεύτερου προγράμματος, την αξιολόγηση και πιο συγκεκριμένα οι αρχές νομοθέτησαν ε, με φιλόδοξες πολιτικές που καλύπτουν πολλούς τομείς της οικονομίας διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις, ενέργεια, ε, εργασιακά. Και το Eurogroup από τη δικιά του την πλευρά ε, παρουσίασε την δικιά του προσέγγιση για την βιωσιμότητα και εγκρίθηκε με 8,5 δισεκατομμύρια συνολικά. Το IMF e επίσης τον Ιούλιο ενέκρινε τους νέους διακανονισμούς και τις αρχές όσον αφορά την Ελλάδα. Όλες αυτές οι θετικές εξελίξεις οδήγησαν σε μια βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά τις αγορές και για πρώτη φορά από το 2014 μπορεί να βγει σε αγορές η Ελλάδα και έχουμε λόγους να είμαστε αισιόδοξοι για την τρίτη αξιολόγηση η οποία γίνεται τώρα όσον αφορά το υπόλοιπο πρόγραμμα. Σήμερα θέλω πρώτα απ' όλα να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις για το πρόγραμμα πριν περάσω πιο συγκεκριμένα στα εργασιακά και θα εξηγήσω πώς οι χώρες μέλη ε, στηρίζουν τις διαδικασίες μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Από τότε που συνελήφθη στο μυαλό μας το πρόγραμμα αυτό για την Ελλάδα, ε, ήθελε να λάβει υπόψη όλα τα επιτεύγματα που γίνονται όσο περνάει ο καιρός και έτσι να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον, όπως είπατε και εσείς ε, κυρία Πρόεδρε. Αυτό θέλουμε και όλοι. Ένα καλύτερο μέλλον το οποίο χτίζεται σε στέρεα θεμέλια. Και όπως ε, μάθαμε τα χρόνια της κρίσης ή από την αρχή από την κρίση, δεν πρέπει να κάνουμε υποθέσεις αβάσιμες, γιατί αυτές οδηγούν στην καταστροφή. 21% ανεργία για τους νέους 40% μερικές φορές. Όλα αυτά ευτυχώς τώρα πάνε κάπως καλύτερα. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε σήμερα δείχνουν ότι η κατάσταση φυσικά εξακολουθεί να είναι απαράδεκτη και χρειάζεται δράση παρά τις όποιες βελτιώσεις. Η βελτίωση λοιπόν της ε, απασχόλησης ε, πάει χέρι-χέρι με μια στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ελλάδα χρειάζεται λοιπόν ένα καλό μοντέλο για επενδύσεις προκειμένου οι επενδυτές να έχουν ε, εμπιστοσύνη. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι κάτι πολύ βασικό ε, για να μπορέσει και η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει το δυναμικό που διαθέτει και το οποίο δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται σήμερα. Ε, χρειάζεται βελτίωση λοιπόν του γενικού πλαισίου για την ανάπτυξη και αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο δουλεύει η Ελλάδα και εμείς και θα συνεχίσουμε. Ο κοινό μας στόχος ήταν έτσι κι αλλιώ να υπάρξει μια καλή εξισορρόπηση για την ανάπτυξη υπέρ της οικονομίας έτσι ώστε όλοι να μπορούν να προσφέρουν ένα καλύτερο και πιο σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Χρειάζονται πόροι για την όσο γίνεται καλύτερη χρήση και κυρίως προς την κατεύθυνση των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας. Και αυτό είναι κάτι που το δουλεύει η Ελλάδα και θα συνεχίσει εφόσον έχει κατακαιρματιστεί το κοινωνικό σύστημα προστασίας στην Ελλάδα. Πρόσφατα η Ελλάδα υιοθέτησε πολλές εργασικές μεταρρυθμίσεις έγινε η πρώτη αξιολόγηση το 2015 που υπο... υπενθύμησε ότι ε, μετά την ε, κρίση χρειάζεται βελτίωση πολλών ε, στοιχείων. Πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική η οικονομία, πιο ευέλικτη για να μπορεί να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά τους πόρους και να διορθωθούν οι ανισορροπίες που είχαν συσσωρευτεί. Η μεταρρύθμιση όμως αγοράς εργασίας φυσικά είναι κάτι πάρα πολύ λεπτό και ευαίσθητο. Κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με μια εύθραυστη ανάκαμψη. Από τη μια μεριά λοιπόν υπάρχει το θέμα του σεβασμού και της ε, τήρησης των κοινωνικών δικαιωμένων των εργαζομένων, από την άλλη μεριά υπάρχει ανάγκη να διατηρηθεί η ευελιξία και να βελτιωθεί η, η ελκυστικότητα της ε, αγοράς. Το θέμα των εργασιακών λοιπόν και οι δυσκολίες αυτές δεν είναι κάτι που μπορεί να αγνοηθεί. Πιστεύω συνολικά ότι οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν ε, μέχρι σήμερα είναι ένας καλό ε, συμβιβασμό μεταξύ αυτών που σας ανέφερα. Πρώτον υπάρχει το πρόγραμμα δράσης τη κυβέρνηση με μέτρα για να αντιμετωπιστεί αδήλωτη εργασία και δεσμεύτηκαν για απλοποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Δεύτερον, σε σχέση με τις συστάσει της ομάδας ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, συμφώνησαν να ξεχρονίσουν ε, τα εργασιακά πλαίσια σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες πρακτικές. Κατά τη γνώμη μου η συμφωνία αυτή βοηθάει στον εξυγχρονισμό της ε, μεταρρύθμισης των συλλογικών συμβάσεων μετά την επιτυχή έκβαση του προγράμματος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ σημαντικό για την ελληνική κυβέρνηση. Όπως και ο εξυγχρονισμός ε, για τις απολύσεις, για τις απεργίες και οι αρχές έχουν ήδη αναλάβει νομοθετικό ε, πλαίσιο από αυτού. Τώρα για την τρίτη αξιολόγηση. Χρειάζεται νομοθεσία ώστε να φανεί ότι λαμβάνουμε υπόψη μας το ποσό το 50% των ε, όσων συμμετέχουν στις δικαλιστικές αποφάσεις. Έπειτα, οι πολιτικές για την βελτίωση της απασχολησιμότητας ε, των ε, ανέργων. Είναι κάτι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της μεταρρύθμισης των εργασιακών. Πρέπει να ενισχυθούν τα επεκτατικά μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να ισχύουν το 2019 και να υπάρχει και βελτίωση της ε, εγγύησης του ελάχιστου εισοδήματος. Έτσι φτάνω στις αποφάσεις που πήρε το Eurogroup στις 15 Ιουνίου για να στηρίξει την ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Πρώτον, συμφωνήσαμε να μειώσουμε την περίοδο κατά την ε, ε, οποία ισχύει το πρόγραμμα 2018 είναι για πέντε χρόνια, δηλαδή μετά το 2022 η Ελλάδα φέχει ένα συνεπές με το ευρωπαϊκό φορολογικό πλαίσιο, ειδικό της πλαίσιο. Δεύτερον, το κύριο Κρόπη βεβαίωσε ε, το θέμα του χρέους και ήδη υπάρχουν μέτρα τα οποία εφαρμόζονται όσον αφορά το έλλειμμα. Και έπειτα υπάρχουν και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν είτε συγχρόνως ή μετά την επιτυχία έκβαση του προγράμματος που προβλέπεται για του χρόνου. Τώρα το Eurogroup φυσικά και τα παίρνει πάρα πολύ σοβαρό όλα αυτά, γι' αυτό και μιλήσαμε για μεσοπρόθεσμα μέτρα όσον αφορά το χρέος. Συμφώνησε το Eurogroup να στηρίξει την Ελλάδα προκειμένου να έχει πρόσβαση στις αγορές, ε, ανακουφίσοντας το χρέος της χώρας αλλά και προκειμένου να δοθούν επιπλέον χρήματα από τον ESM μετά την ε, περίοδο του προγράμματο. Και θα ολοκληρώσω λέγοντα ότι οι αποφάσει οι οποίε έχουν ληφθεί μέχρι τώρα βάσει του προγράμματο του ESM βασίζονται στα αποτελέσματα ε, τη Ελλάδα και στην πρώτη ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει με τι μεταρρυθμίσει. Και το Eurogroup αποφάσισε να στηρίξει την Ελλάδα στη διαδικασία αυτή, επιδεικνύοντα παρετέρω αλληλεγγύη. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά βέβαια του επόμενου μήνε και χρόνια. Το Eurogroup ενθαρρύνει την Ελλάδα να συνεχίσει να δουλεύει υπέρ μια μακροχρόνιας αξιόπιστης ανάπτυξη σε συνεργασία με του εταίρου. Το τρίτο πρόγραμμα, η εξολόγηση μάλλον του τρίτου προγράμματο, γίνεται αυτή την εποχή, γίνονται συζητήσει ανάμεσα στου θεσμού και τι αρχέ. και το πνεύμα είναι ιδιαίτερα επικοδομητικό. Είμαι βέβαιο ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την τρίτη αυτή αξιολόγηση μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Και αυτό είναι κάτι που θα επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα έχει μπει στο σωστό δρόμο ε, και θα βγει από το πρόγραμμα επιτυχώς την επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στους συντονιστές ξεκινώντας από τον κύριο Μπέκερ που ε, εκπροσωπεί τον κύριο Κάζα. Παρακαλώ. Ähm, äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ως ε, υποσυντονιστής του ΕΛΚ θα ήθελα να επενέσω τη δουλειά του Eurogroup ε, όσον αφορά την Ελλάδα. Βλέπουμε και τους πρώτους καρπούς. Ε, βλέπουμε θετικά στοιχεία ε, όσον αφορά τα επιμέρους κριτήρια. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι το ΕΛΚ ε, επικροτεί την σωστή εφαρμογή του προγράμματος από την ελληνική κυβέρνηση Θέλουμε όμως να τονίσουμε ότι στο μέλλον αυτό δεν θα πρέπει να αλλάξει στο μέλλον, θα πρέπει να ενταθεί, διότι ακόμα δεν έχει διασφαλιστεί ο στόχος ενός διασφαλισμένου μέλλοντος. Όσον αφορά την οικονομία, η ανάπτυξη δείχνει πόσο μακροπρόθεσμα είναι τα μέτρα του Eurogroup. Η οικονομική ανάπτυξη αναθεωρήθηκε κατά 0,6%. Ποιοι είναι οι λόγοι για κάτι τέτοιο. Τρίτον, η Ελλάδα από τον Ιούλιο του 2017 συμμετέχει πάλι στις, οικονομικ... στις Ε, και μάλιστα με πολύ θετικά αποτελέσματα. Το Eurogroup πώς θα εκμεταλλευτεί αυτά τα αποτελέσματα. Ε, πρέπει ε, να καταπολεμηθεί η ανεργία στην Ελλάδα αποτελεσματικά. Πώς το βλέπει αυτό το Eurogroup. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Then I'll give the... Ευχαριστώ κύριε Μπέκερ. Δίνω το λόγο στην κυρία Γιονγκέριου, σε συντονίστρια του S&D. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Γερούν που είσαι παρόν εδώ στην Επιτροπή μας. Θα αναφερθώ σε κάτι που μας ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτερα. Όχι μόνο το πώς θα πηγαίνει η οικονομία στην Ελλάδα, αλλά και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους απλούς εργαζομένους στην Ελλάδα και τους ανθρώπους που, που εξαρτώνται από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Να πω καταρχάς ότι κατά τη γνώμη μας ε, το αίτημα για την αποκατάσταση των ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα είναι η κορυφαία, κορυφαία, κορυφαία προτεραιότητά μας. μετά την τρίτη αναθεώρηση του προγράμματος. Είπες ότι θα, μπορέσει, θα μπορέσουν να γίνουν διαπραγματεύσεις για ένα εξυγχρονισμένο σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ελπίζω, αλλά ίσως να μπορείς να μας διαφωτίσεις. Νομίζω ότι διαφωνούμε όσον αφορά το κατά πόσο το ισχύον σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανόνες του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το ε, Συμβούλιο της Ευρώπης έχει κρίνει παράνομο, τη, παράνομη την ε, μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας από την Τρόικα. Και το ILO, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, επισημαίνει τον περιορισμό της κάλυψης ε, των Ελλήνων ε, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Μπορείς λοιπόν να μας πεις τι γίνεται όσον αφορά το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων, πότε θα εφαρμοστούν όλα αυτά και κατά πόσο θα συνάδουν με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και κατά πόσο θα μετριαστούν τα προγράμματα που εμφανίστηκαν μετά την αναθεώρηση του 2015. Ευχαριστώ. Ε, okay, we'll go to... Καλώς λέει Πρόεδρος. Και τώρα για την ECR. Η κυρία Μακιντάιρ, αλλά απουσιάζει. Α, όχι, όχι, εδώ είναι, εδώ είναι. Α, ντυμένη τόσο ωραία, μέσα στα ροζ. Και δεν σας είδα παρόλα αυτά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ήξερα ότι ήμουν αόρατη και ξαφνικά με είδατε. Εκπροσωπώ χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωζώνη. Μια χώρα που μπόρεσε ευτυχώς να συρρυκνώσει τα ποσοστά της ε, ανεργίας ε, σε σημείο ρεκόρ. Τώρα δημιουργούμε θέσεις ε, απασχόλησης επί κάποια έτη. Και είναι κάποιες θέσεις εργασίας που φτιάχνουμε που κατά τα τρία τέταρτα είναι μόνιμες. Δεν, δεν είναι μερική απασχόληση. Δεν είναι για βραχυπρόθεσμη απασχόληση. Θα ήθελα να δούμε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό είναι το εξής. Να επικεντρωθούμε στις δεξιότητες. Ξέρουμε ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει έλλειψη κάποιων δεξιοτήτων όπως ε, ε φυσικές επιστήμες ε, και όχι μόνο. Οπότε, όπου υπάρχουν τέτοιες δεξιότητες πρόκειται να γίνουν οι επενδύσεις. Αυτό τις ελκύει τις επενδύσεις. Άρα απλά απασχόλησης με ενδιαφέρει να μου πείτε τι κάνει η Ελλάδα πάνω σε αυτό. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί σε απασχόλησης. Έτσι. Και όχι με τον άλλο τρόπο που βέβαια και αυτός είναι σημαντικός. Και έτσι να μπορέσουμε για να περιστύλουμε την μαύρη εργασία. Μόλις τώρα είπαμε με την πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδειλωτής εργασίας. Οπότε θέλω να ξέρω και η Ελλάδα ωφελήθηκε από την πλατφόρμα για καταπολέμηση άτυπης εργασίας. Επίσης, ε, διαβάζω ότι μέχρι 20% της ε, οικονομικής δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι στην παραοικονομία με την αδίλωτη εργασία και σε μερικού τομείς πάμε στο 40%. Αυτό το νούμερο μου φαίνεται τερατώδη στη δική μας ε, χώρα. Είμαστε στο 1,7%. Επομένως υπάρχει τεράστιο περιθώριο βελτίωσης και δεν όλα με τη δίωξη και με τα δικαστήρια παρά το ότι έχουν παρανομήσει αλλά ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούσαμε προηγουμένως δηλαδή πως ενθαρρύνουμε κάποιον να νομιμοποιηθεί να μπει από την μαύρη στην κανονική οικονομία αυτό, αυτό με ενδιαφέρει να ακούσω από εσά. Ο κύριος Καλβέτ Τσαμπον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Ντάσελμπλουμ. Θα είμαι σύντομο. Πρώτα πρώτα. Μια που συζητούμε για την Ελλάδα είχε και έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Δεν έχει κάποιες βασικές οικονομικές δομές. Ούτως ώστε πραγματικά να μπορέσουν να εξασφαλίσουν κάποια επαρκή διαχείριση της οικονομίας. Όλα αυτά τα πήγαιναν στην Ευρωζώνη. Δεν είχε η Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχει τώρα, ένα φορολογικό σύστημα σοβαρό, αντίστοιχο με τις υπόλοιπες δυτικές χώρες. Οπότε, για πιστεύω μου τη γνώμη σας. Αν αναπόφευκτα θα πρέπει να γίνουν κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί από κάποιο είδου κοινωνική απορρόφηση. Λογική. Δηλαδή να μην πάμε με τις μεταρρυθμίσεις αυτές τις διορθωτικές να καταλήξουμε σε ένα νεκροταφείο της απασχόλησης. Και εδώ είναι η σημαντική ερώτηση. Μπας και οι ελληνικές αρχές βάζουν τροχοπέδια ή υπάρχει τέλο πάντων κάποιος φραγμός. συμπαθώντα με για το τηλέφωνο, το, το κλείσα. Βάζουν λοιπόν τροχοπέδια στα μέτρα. Δηλαδή δεν πιστεύουν σε αυτά τα μέτρα ή δεν πιστεύουν ότι είναι απαραίτητα για τον εξυγχρονισμό της ε, χώρας. Και έτσι δεν μπορεί να εφαρμοστεί τίποτα. Αυτό ήταν η μια ερώτηση. Δεύτερον, κύριε Ντάσελμπλουμ. Οφείλω να σας πω ότι το ευρώ έχει νόημα μόνο και αποκλειστικά εάν δίνει ευημερία σε όλους τους Ευρωπαίους. Τους κάνει πιο ελεύθερους. Τους προστατεύει περισσότερο. Να μην αποτελεί στα χέρια των τραπεζιτών. Είναι ένα εργαλείο πολύ σημαντικό για την κοινωνική ευημερία. Ε, σε αυτό θα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει για να πείσουμε περί τούτου τους Ευρωπαίους. Εκεί η δική μου χώρα βέβαια φύγει πάρα πολύ από την ε, κρίση. Προέχουμε μία από τις χώρες εκείνες που είπατε ε, αυτό τους συμβαίνει γιατί αυτό το οποίο κάνουν είναι να τα πίνουν και να τα ξοδεύουν στις γυναίκες. Ε, ναι, αλλά έτσι όμως αυτό το οποίο κάνετε είναι να δημιουργείτε άρνηση προς το ευρώ ε, θα έπρεπε να δημιουργείται ένα θετικό κλίμα, ένα ευμενές ε, προς το, τον απλό κόσμο, τον απλό κόσμο που δεν είναι μεγάλος οικονομολόγος όπως εσείς. Α, δεν έχω χρόνο να Λοιπόν, εσείς θα πρέπει να συμμετάσχετε σε κάποιο διαπαιδαγώγηση του κόσμου και να μάθετε στον κόσμο ότι πρόκειται το ευρώ να είναι εργαλείο για να τους φέρει ευτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Παπαδημούλης. Sorry. Ε, Κύριος Χουντής, συγγνώμη, διορθώνει πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κύριε Ντάζερμπλουμ, εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, είμαι Έλληνας Ευρωβουλευτής, διότι η δική συζήτηση με εσάς, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, είναι η πιο αυθεντική σχετικά με το πώς πάνε τα μνημόνια και ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω από την ώρα που συγκροτήθηκαν και επευλήθηκαν τα μνημόνια στην Ελλάδα υπήρχε ένας διάλογος στο δημόσιο τομέα ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ζητάτε μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχία, ενώ μεταρρυθμίσεις και κυρίως τα εργασιακά με στόχο την υποβάθμιση της εργασίας και της κοινωνίας τα ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ερώτηση πρώτη. Είναι αληθές αυτό. Ερώτηση δεύτερη η πορεία έδειξε ότι μέσα στα μνημόνια και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δέχτηκαν να υπάρχουν και τέτοια μέτρα. Ερώτηση. Ισχύει τελικά ο χάρτης θεμελιδών δικαιωμάτων για χώρες που είναι στο πρόγραμμα, διότι έχω πάρει αντιφατικές απαντήσεις. Ο κύριος Γιούγκερ λέει όχι. Η αρμόδια Επίτροπος Επικοινωνικών Υποθέσεων πρόσφατη ερώτηση λέει όχι και το τηρούμε. Τρίτη ερώτηση. Αυτά τα μέτρα για τις συλλογικές συμβάσεις για τις ομαδικές απολύσεις, για τα ε, επιπτώματα που κόβονται, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ισχυρίζονται ότι τα ζητάει και τα προτείνει η ελληνική κυβέρνηση. Και δεν τα ζητάτε εσείς. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η αλήθεια. Και τέλος, με την ευκαιρία που σας είχα γνωρίσει στην προηγούμενη θητεία όταν, είχα αναλάβει, όταν είχατε αναλάβει για πρώτη φορά ε, την Προεδρία του Eurogroup. Και είσαστε περήφανος διότι εσείς εμπνεύστηκατε ε, το κούρεμα των καταθέσεων των κυπριακών καταθέσεων τότε. Τώρα φεύγετε. Ερώτηση, λοιπόν. Την έκανε ως ένα βαθμό ένα συνάδελφος. Επιμένετε, λοιπόν, ότι οι Έλληνες έπρεπε να τιμωρηθούν, διότι ήταν τεμπέλιδες και σπάταλοι. Επιμένετε ότι αυτά τα προγράμματα ήταν αλληλεγγύη και στήριξη στην Ελλάδα ή θα παραδεχτείτε Πράγμα που έκανε ο κύριος Ρεν, ο προηγούμενος επίτροπος, όταν έφευγε. Ότι αυτά τα προγράμματα ήταν για να στηριχτούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και το ευρώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κούνεβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντάισελμπρουμ, είναι πολύ σημαντικό ο εκπρόσωπος του Eurogroup να βρίσκεται ανάμεσα εδώ, διότι οι κοινωνικές πολιτικές δεν είναι δυνατόν να αποφασιστούν χωρίς τη στήριξη των οικονομικών αρχών. Αυτό το διαλαλούν εδώ και χρόνια οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Για την Ελλάδα όμως είπατε και εσείς η αξιολόγηση πηγαίνει καλά. Φαίνεται να ικανοποιούμε τους δείκτες τους οποίους απαιτείται. Τι γίνεται όμω με τους κοινωνικούς δείκτε. Προτεραιότητα στην απασχόληση δεν πρέπει να δίνουμε μόνο η Επιτροπή απασχόληση, Δεν πρέπει να δίνει μόνο η UTUC, το ΕΤΟΚ, η οποία με έκθεσή τη εχθέ υπογραμμίζει πως η κατώτατη μισθή σε πολλέ χώρε της Ευρωπαϊκή Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, είναι πολύ χαμηλότερη από το αποδεκτό όριο με αποτέλεσμα πολλοί Ευρωπαίοι εργαζόμενοι να μην μπορούν να επιβιώσουν εργαζόμενοι. Προτεραιότητα πρέπει να δίνουν όλοι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θέλουμε να σταματήσουμε την επικίνδυνη αύξηση του λογισμού στην Ευρώπη. Για να ξανακερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών πρέπει να τους επιστρέψουμε την αξιοπρέπειά τους. Και όχι με λόγια, αλλά με έργα. Λέτε πώς στηρίζετε. Πώς ακριβώς όμως. Στην Ελλάδα η συνέπειες της απασχόληση σε συνδυασμό με την κρίση ήταν καταστροφικές. Λέτε για την Επιτροπή των Σοφών και τα εργασιακά. Η Επιτροπή είπε πως η Ελλάδα ήδη ακολουθεί τις καλές πρακτικές. Άρα, εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό. Πρέπει να ακούσουμε αυτή την Επιτροπή. Νομίζω ότι πρέπει να δείτε πιο καλά τι λέει η Επιτροπή των Σοφών. Η Ελλάδα υποβάλλει συγκεκριμένε προτάσει για την τόνωση τη απασχόληση προτείνει η επενδύσεις στην απασχόληση, ειδικά για τους νέους και τους μακροχρόνια άνεργους, να μην συνυπολογίζεται. Είναι μια πρόταση με έντονη στήριξη από τους υπουργούς απασχόλησης της Ευρώπης. Τα προτατήκες τα προτατήκε στον πρόεδρο της Κομισιόν και στους αρμόδιους επιτρόπους. Εσείς στο Eurogroup την έχετε απορρίψει. Μπορείτε να μας πείτε γιατί. Και ποια είναι η αντιπρότασή σας. Και στο τέλος θέλω να εκλυπαρώ να μη σκοτώνει η Eurogroup το κοινωνικό πυλώνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω το λόγο βέβαια και στους ε, υπόλοιπους είτε συντονιστέ είτε οτιδήποτε τόσο πάντων που ζήτησαν το λόγο, αλλά να είσαστε σύντομοι παρακαλώ. Γιατί πρέπει να υπάρχει χρόνος να ακούσουμε και τον κύριο Ντάσελμπλουμ τι έχει να απαντήσει. Έτσι και δεν έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Καλό θα ήταν να μας πείτε και ποιος εκπροσωπεί τις ομάδες όταν δεν υπάρχει εδώ συντονιστής παρόν, να ξέρουμε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κυρία Κούνεβα. Παρακαλώ, σύντομα όμως. Με συγχωρείτε, γίνει λάθος ε, στη μετάφραση. Είπα ότι η, η Επιτροπή των Σοφών έχει πει ότι η Ελλάδα ακολουθεί τις καλές πρακτικές της Ευρώπης ότι η Ελλάδα έχει ακολουθήσει και ακολουθεί τις καλές πρακτικές της Ευρώπης. Το έχει πει η Επιτροπή των Σοφών. Ωραία. Μάρκο Βάλε, παρακαλώ. Σύντομα, πολύ πρόεδρε, όπω και εσείς ε, ζητείτε, υποκαθιστώ την κυρία Ντετζία της ε, EFD που δεν μπορούσε να παραστεί σήμερα. Όσον αφορά τώρα το θέμα των μεταρρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί στις χώρες τη Ευρωζώνη, μα ε, μας, στρίμωξε πάρα πολύ και την Ιταλία και την Πορτογαλία και την Ισπανία και την Ελλάδα και σήμερα κάνατε αυτή την ανάλυση για το ότι η ανάπτυξη οφείλεται ε, κατά πολύ στις ε, μεταρρυθμίσεις. Ναι, αλλά εμείς νομίζουμε ότι αυτή η ανάπτυξη πάσχει σε πολλά σημεία, εξού και τα προβλήματα ρευστότητα σε πολλές ε, τράπεζες και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα, επομένως, που έχουμε κανένα απτό συγκεκριμένο αποτέλεσμα ε, σε σχέση με τα χρήματα τα οποία μπήκανε μέσα στο χρηματοοικονομικό κύκλωμα όσον αφορά δηλαδή την, ε, τον πληθωρισμό, την απασχόληση, τι γίνεται με την ζήτηση η οποία έχει καταρρεύσει. Τι γίνεται με αυτές τις μεταρρυθμίσεις της περιφέρειας της Ευρώπης. Η Ευρωζώνη κατά κάποιο τρόπο θέλει να κάνει αυθεντικές μεταρρυθμίσεις, να μην υπάρχουν εσωτερικές ε, ανισορροπίες, να μην ε, εξευτελιστεί το, η εργασία ε, σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα. Εσείς όμως στη χώρα σας έχετε άλλου είδους κίνητρα, όπως και η Γερμανία με το πλεόνασμά τους θέλουν να κάνουν το δικό τους τρόπο ε, κατανομής του χρέους για την Ιταλία, για την Ελλάδα και τις μεταρρυθμίσεις τις βάζετε και στην περιφέρεια. Θα υπάρχουν όμως κάποιες πολιτικές δυνάμεις οι, οι οποίες με την επόμενη κρίση θα θέλουν να βγάλουν τις χώρες από την Ευρωζώνη. Οπότε νομίζω θα πρέπει αυτή η προβληματική να ισχύσει, να συζητηθεί τέλο πάντων στο Eurogroup. Θα πρέπει να αποδεχθούν κάποια πράγματα οι χώρες Βόρειας Ευρώπης. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω τον κύριο Χουντή στον κατάλογο και τον κύριο Παπαδημούλη. Δεν θέλετε να πάρετε το λόγο. Uh, and then we have Και έχουμε την κυρία Ρέγνερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι σοσιαλδημοκράτρια από την Αυστρία και έχω δύο ερωτήσεις, κύριε Ντάισλμπλουμ. Καταρχάς, θεμελιώδη δικαιώματα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι θεμελιώδη δικαιώματα εξορισμού. Ε, το δικαίωμα απεργίας, το δικαίωμα ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων πρέπει να γίνονται σεβαστά και σε, και σε καλούς και σε δύσκολους καιρούς. Αναφερθήκατε στις εξυγχρονισμένες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Μπορείτε να μας πείτε τι μορφή θα έχουν, ε, έχοντας υπόψη ότι μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα. Δεύτερον, όσον αφορά τη συζήτηση για τις δεξιότητες στο Eurogroup. Όλοι γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε ε, θέσεις απασχόλησης υψηλών δεξιοτήτων ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. Τώρα, όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα, όταν βλέπουμε λίγο φως στην άκρη του τούνελ, βλέπουμε ότι η παραγωγή δεν ε, αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν θέσεις εργασίας ε, χαμηλής αμοιβή και χαμηλών δεξιοτήτων. Αυτό λοιπόν ε, θα είναι το μέλλον για την Ελλάδα, να είναι ανταγωνιστική με αυτές τις ε, θέσεις απασχόλησης χαμηλών δεξιοτήτων. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσει αυτήν την οδό. Και με ενδιαφέρει να ακούσω όχι μόνο το πώς συζητιέται, αλλά και ποια είναι η δική σας προσέγγιση στο Eurogroup. Ποια είναι η πραγματικότητα και ποιες είναι οι επιθυμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ο κύριος Ροχφόρτ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Κύριε Ντάσελμπλουμ, σίγουρα μετράνε οι πολιτικές, αλλά από τη δικιά σας την πλευρά, από τη θέση στην οποία βρισκόσαστε, πρέπει να κοιτάτε και την οικονομική πραγματικότητα, το πώς έχουν τα πράγματα, λέτε, οικονομικά. Και Πολύ προβληματίζομαι από την αρχή τη συζήτηση για το κατά πόσο υπάρχουν πραγματικά αποτελέσματα στην Ελλάδα σήμερα. Οι προβλέψει ανάπτυξη για το 2015 να θεωρούνται προ τα κάτω. Η ανάπτυξη που θα έπρεπε να είναι κάπω θετική το 2016, αν δούμε τη δεύτερη εκτίμηση, είναι αρνητική. Και μιλάμε και για την ανεργία και λέμε ότι μειώνεται. 23 με 21,5% είναι σημαντική αυτή η μείωση. Σήμερα στην Ελλάδα φαίνεται ότι έχουμε διαρροές ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι καταλείπουν τη χώρα και οι οποίοι όμως είναι υψηλών προσόντων. Συχνά μιλάμε για την ανεργία των ανεδίκευτων, αυτών που είναι λιγότερο παραγωγή κτλ. όπως είπε συνάδελφος πριν, αλλά εμένα αυτό που ανησυχεί ακόμα πιο πολύ είναι ότι φεύγουν διαρροή εγκεφάλων, ότι φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα, οι οποίοι εκπαιδεύονται για να ηγηθούν μιας παραγωγικής οικονομίας και θα έπρεπε να το κάνουν αυτό στην Ελλάδα, όπου δεν μπορεί να είναι μόνο τουρισμό η πηγή πλούτου, θα έπρεπε να υπάρχει παραγωγή. Αν λοιπόν δεν πάμε πιο γρήγορα, αν δεν έχουμε προγράμματα επενδυτικά ε, περισσότερο στρατηγική σημασία και πιο ισχυρά, μεθαύριο η Ελλάδα θα είναι μια χώρα όπου εκατοντάδε χιλιάδε νέοι που έχουν εκποδοθεί, μιλάμε ήδη για ε, πάρα πολλού που φύγανε τα τελευταία χρόνια, θα λείπουν από τη χώρα. Πώς θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα λοιπόν η Ελλάδα μέσα σε αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Παπαδημούλης τώρα τελικά θέλει να ρωτήσει κάτι. Ε, δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο. Ήρθα να ακούσω τον κύριο Ντάισελμπλουμ γιατί τα συζητάμε συχνά και στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια και στην ειδική ομάδα εργασίας που έχει συγκροτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρακολουθεί κοινοβουλευτικά την εξέλιξη της εφαρμογής του τρίτου προγράμματος. Ζήτησα το λόγο για να πω σε όλους τους συναδέλφους όλου του φάσματος ότι σήμερα έδωσε η Κομισιόν τις εκτιμήσεις της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας που λένε ότι η Ελλάδα έχει επιστρέψει μετά από χρόνια ύφεσης και οδυνηρών θυσιών του ελληνικού λαού σε μια τροχιά ανάπτυξης. Προβλέπει μια ανάπτυξη 1,6% για φέτος, 2,5% για το 2018 και 2,5% για το 2019. Η ανεργία παραμένει υψηλή, αλλά πριν δύο χρόνια ήταν 27% και τώρα είναι 21% η ανεργία των νέων παραμένει πολύ υψηλή, είναι στο 40% όπως είπε ο κ. Ντάισελουμ, αλλά πριν δύο χρόνια ήταν στο 55% και όλο ένα και περισσότεροι παράγοντες και ο κύριος Ντάισελμπλουμ και ο κύριος Ρέκλινγκ και η Κομισιόν εκτιμούν ότι είναι εφικτό η χώρα μου να βγει από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε πάρα πολύ τις συνέπειες μιας κακής διακυβέρνησης για χρόνια στο παρελθόν που προκάλεσε ελλείμματα και χρέη, αλλά και λάθος συνταγές που προκάλεσαν τεράστια ύφεση, τεράστιο κοινωνικό πόνο, τριπλασιασμό της ανεργίας, έχουν αρχίσει να δημιουργούνται κάποια φύτρα θετικά, αρχίζουν να παράγονται πια και κάποιες θετικές ενδείξεις. Αυτό είναι το μήνυμα που πήρα εγώ από τον κύριο Ντάισεμπλου, με τον οποίο έχουμε διαφωνήσει έντονα πολλές φορές στο παρελθόν. Και θα ήθελα να πω ότι αυτή την ώρα, αν κάτι πρέπει να κάνουν όλες οι πλευρές, και η ελληνική κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι δανειστές και οι εκπρόσωποι των θεσμών, είναι να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης για να τελειώσουμε το συντομότερο δυνατό ή δυνατόν να έχουμε staff level agreement το Δεκέμβριο και θα ήθελα σε αυτό να ρωτήσω τον κύριο μου ποια είναι η εκτίμησή του, έτσι ώστε το πρώτο εξάμεινο του 2018 να σχεδιαστεί το phasing out από το πρόγραμμα, να συγκεκριμενοποιηθούν τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που αποφάσισε το του 15 Ιουνίου και να μπορέσει η Ελλάδα να βγει οριστικά από αυτήν την εντατική θεραπεία της μηχανικής υποστήριξης που σημαίνει μνημόνια για να αποκτήσουμε και πάλι τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και όλοι οι λαοί που επιλέγουν να είναι στην Ευρωζώνη. Αυτό ήθελα να πω, γιατί νομίζω ότι ορισμένες τοποθετήσεις συναδέλφων έχουν μείνει ένα-δύο χρόνια πίσω σε σχέση με τις εξέλιξεις. Ευχαριστούμε. Κύριε Ντάσελμπλουμ, έχετε 20 λεπτά στη διάθεσή σας, παρακαλώ, για να απαντήσετε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Χωρίς βέβαια να θέλουμε και να σας τρεσάρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ όλους τους αξιότιμους ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Έχετε δίκιο να είσαστε επικριτικοί και έχετε δίκιο να προβληματίζεστε για το μέχρι τώρα έργο μας. Παρ' όλα αυτά, έχουμε περάσει σε ένα επόμενο στάδιο Υπενθυμίσατε πολύ από εσά τα στοιχεία και λέτε ότι αναθεωρούνται προς τα κάτω. Ε, Παρ' όλα αυτά, σε σχέση με την περσινή κατάσταση, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σήμερα. Ναι, η εκτίμηση της ε, Επιτροπής ήταν πιο φιλόδοξη, ήταν ε, πιο αισιόδοξη μάλλον, 2,1%. Τώρα φαίνεται ότι είμαστε στο 1,6%. Αλλά πριν δεν υπήρχε καθόλου ανάπτυξη. Οπότε υπάρχει πραγματική βελτίωση. Έχετε δίκιο ότι η ανεργία βρίσκεται σε επίπεδα παράδεκτα ακόμα. Και πιστεύω ότι η εκτίμηση για φέτος θα είναι 21%. Πριν από τέσσερα χρόνια ήμασταν στο 28%. Οπότε υπάρχει πραγματική βελτίωση. Ε, φτάνει? Όχι βέβαια, κάθε άλλο. Και γι' αυτό και επιμένουμε σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και με και όλοι οι θεσμοί της κυβέρνησης έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες και μπράβο τους που προσπαθούν να βελτιώσουν και την καθημερινότητα των ανθρώπων και τις προοπτικές κυρίως των νέων. Το θέμα της ανεργίας είναι πραγματικά τρομερό. Οι μεταρρυθμίσεις τώρα που έγιναν και ρωτήσατε για το χρονοδιάγραμμα αν είναι μακροπρόθεσμες και αν θα παραμείνουν μετά το τέλος του προγράμματος. Εντάξει, κάποια στιγμή θα υπάρξει το τέλος του προγράμματος, σίγουρα την επόμενη χρονιά. Από εκεί και πέρα είναι στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Βάσει των συμφωνιών που έχουμε στην Ομισματική Ένωση να φροντίσουν για την δημοσιονομική βιωσιμότητα, για τις καθημερινές βελτιώσεις στην αγορά εργασίας, στην παραγωγικότητα, να, βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι προδιαγραφές στην εκπαίδευση κλπ. κλπ. Είναι μια βασική στιγμή. Αύγουστο λύγει το πρόγραμμα και από εκεί και πέρα η Ελλάδα στέκεται μόνη στα πόδια της, όχι μόνο δημοσιονομικά, αλλά και όσον αφορά τις πολιτικές που θα υιοθετεί. Δεν υπάρχει βέβαια θέμα ανατροπής των μεταρρυθμίσεων, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες, να υπάρχει συνεχής προσπάθεια για βελτίωση. Αναφερθήκατε και στην πρόσβαση στις αγορές. Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα. Η Ελλάδα πριν από λίγους μήνες βγήκε στις αγορές και θα συνεχίσει να το κάνει δοκιμάζοντας τις ε, αγορές κάθε τόσο. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να πηγαίνει συχνά τα επόμενα χρόνια στις αγορές, δεδομένου ότι έχουν πρωτογενές πλεόνεσμα, ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι είναι πάνω από τους ε, βασικούς στόχους. Οπότε υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για να βελτιωθούν οι κοινωνικές προδιαγραφές με τα στόδομα στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι και θα είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση στην Ελλάδα. Είναι θέμα βέβαια εμπιστοσύνης και βάσει αυτής θα μπορέσει να γίνει πλήρως ανεξάρτητη η Ελλάδα. Δεν υπάρχει, θέλω να πω, σοβαρός λόγος να θέλει η Ελλάδα να βγαίνει στις αγορές. Δεν υπάρχει ανάγκη και αυτό είναι θετικό. Τώρα πολλοί από εσά αναφερθήκανε στα μέτρα για την μείωση της ανεργίας και τις προσπάθειες που έγιναν. Είναι μέρος του προγράμματος η βελτίωση των πολιτικών ε, στην αγορά εργασίας, ακριβώς για να υπάρξει βελτίωση στην επαγγελματική κατάρτιση, Όλα αυτά είναι μέρος του προγράμματος. Τεχνική αρρωγή υπάρχει ακριβώς για να ενεργοποιηθούν ακόμα περισσότερο πολιτικές υπέρ της απασχόλησης. Στήριξη από το Κοινωνικό Ταμείο επίσης υπάρχει και διάφορα προγράμματα στήριξης της αγοράς. Όλα αυτά γίνονται με μεγάλη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων θεσμών για να στηριχτεί η Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια. Είναι κάτι που δεν προβάλλεται τόσο πολύ. Ε, συχνά τα θετικά δεν προβάλλονται αρκετά. Υπάρχουν όμως. Γίνεται πολλή δουλειά και από αυτού. Η κυρία Γιονκέριους αναφέρθηκε στις συλλογικέ ε, συμβάσεις και λέει ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Εντάξει, ερχόμαστε από την ίδια παράδοση ε, σοσιαλδημοκράτες ε, της Ολλανδίας είμαστε και δύο, το σύστημα των συλλογικών συμβάσεων βασίστηκε τουλάχιστον το οριζόντιο σκέλος πάγωσε. Και αυτό είχε να κάνει με την ανάγκη να διορθωθεί η μεγάλη άνοδος στους μισθούς που είχε παρατηρηθεί. Ήταν βέβαια καταστροφικό για την ατοχή της ε, ελληνικής οικονομίας. Αν δείτε, οι μισθοί στην Ελλάδα πώς ανέβηκαν από τη στιγμή που εισήχθη το ευρώ μέχρι την αρχή της κρίσης, ήταν πολύ μεγαλύτερη άνοδος αυτή από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. 30%. Τώρα βέβαια έχει διορθωθεί αυτό και φυσικά οι επιπτώσεις οικονομικές και κοινωνικές είναι αρνητικές. Αλλά έγινε αυτή η διόρθωση σε σχέση με τα χρόνια πριν την κρίση που οδήγησαν στο διέξοδο. Βέβαια, η επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων αποτελεί προτεραιότητα και θα ισχύσει στα τέλη του προγράμματος. Κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη χρονιά δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό. Όταν μιλάμε τώρα για ένα εξυγχωρισμένο σύστημα, σύγχρονο σύστημα, εννοούμε την αντιπροσωπευτικότητα των μερών που συμμετέχουν στις συλλογικέ συμβάσει. Η Ελλάδα έχει ένα κανόνα που λέει ότι πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές οι συλλογικέ συμβάσει. Αλλά ε, δεν ξέρουμε αν αυτό συνέβαινε όντω ή όχι. Τώρα λοιπόν δημιουργείται ένα σύστημα προκειμένου να υπάρχουν τα δεδομένα και να είναι ε, σίγουρο ότι όταν υπάρχει συλλογική σύμβαση σε κάποιο κλάδο, τηρεί και τα κριτήρια της αντιπροσωπευτικότητας. Και άρα ε, μπορεί να έχει δεσμευτικό οριζόντιο χαρακτήρα. Πάνω σε αυτό το στοιχείο δουλεύουμε και αυτό πρέπει να ισχύσει. Και αυτό εννοώ όταν μιλάω για ένα σύγχρονο σύστημα. Και εδώ βέβαια έρχομαι και στο πιο βασικό θέμα γενικώ των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων που ρωτάτε εφαρμόζονται στο πρόγραμμα. Εφόσον το πρόγραμμα διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, πρέπει. Κάποιος από εσά είπε ότι η Επιτροπή δεν ήταν σαφής πάνω σε αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ ασαφής η Επιτροπή από αυτού είναι υπεύθυνη εν μέρη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, οπότε προφανώς και πρέπει να εφαρμόζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και να τα σέβεται. Οι επιπτώσεις της κρίση όμως είναι υπαρκτέ, είναι πραγματικές και χρειάζονταν διορθώσεις για να βγούμε από την κρίση. Και αυτό βέβαια έχει επιπτώσει στον κόσμο. Τώρα, για τις δεξιότητες τα ΕΠΑ. Ήδη είπα για τη συμμετοχή τεχνική αρρωγή της Κομισιόν και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έρχομαι τώρα. κυρία Μακαντάιρ, ρώτησε για την αδήλωτη εργασία που είναι μεγάλη. Είναι πράγματι πρόβλημα. Και έχει να κάνει με τη λειτουργία των θεσμών. Αν λειτουργεί καλά το φορολογικό, ε, μπορεί να αντιμετωπιστεί η αδήλωτη εργασία σε έναν βαθμό. Οι φόροι είναι πολύ ψηλοί στην Ελλάδα ακόμα. Προκειμένου να υπάρξει επανεσυσορρόπηση του δημοσιονομικού, οι φόροι είναι υψηλοί, που φυσικά και έχουν αρνητικέ επιπτώσει, γιατί αυτό σημαίνει ότι ακόμα περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να φοροαποφύγουν. Πώ θα το διορθώσουμε, με τον καιρό. Να έχουμε μια πιο ελκυστική οικονομία και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους, να υπάρχουν οι καταληθεσμοί οι οποίοι θα πιέζουν προς τη σωστή κατεύθυνση, να πληρώνουν δηλαδή ό,τι πρέπει να πληρώνουν και εργοδότες και εργοζόμενοι μέσα σε μια επίσημη οικονομία και όχι άτυπη. Ο κύριος ε, Σαρλίτ Σαμπών αναφέρθηκε σε άλλες ελληνικές αρχές αν συνεργάζονται ή παρεμποδίζουν. Οι ελληνικές ε, αρχές, ξέρετε, το καλοκαίρι του 2015 θυμόσαστε την τεράστια κρίση από την οποία περάσαμε και όπου η εμπιστοσύνη ήταν στο Αδύρ. Όμως, από τότε ε, προχωρήσαμε. Είμαστε σε νέα συμφωνία και έκτοτε η συνεργασία ήταν ε, καλή. Οπότε είμαι θετικός και η δεύτερη αξιολόγηση ίσως εντάξει, πήρε υπερβολικά πολύ χρόνο κάτι το οποίο εμπόδισε την οικονομική ανάκαμψη. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι σήμερα. Τα προγράμματα, οι αξιολογήσει, ε, οι θεσμοί κυριαρχούν, ναι, το ξέρω. Και αυτό επηρεάζει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Αν το πρόγραμμα πηγαίνει καλά, αν η αξιολόγηση τρίτη προχωρήσει ήπια, εύκολα και όντω ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη τη χρονιά, αυτό θα τροφοδοτήσει εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Και θα νιώσουν όλοι ότι κάτι πάει καλά εκεί. Και γι' αυτό είμαι πολύ ικανοποιημένο από τις επικοδομητικές συζητήσεις που έχουμε τώρα με την ελληνική κυβέρνηση και από το γεγονός ότι η τρίτη αξιολόγηση πάει τόσο καλά. Πολύ σημαντικό για να πετύχουμε αυτή την ανάπτυξη του χρόνου. Κάποιος είπε ότι η εκτίμηση ήταν 2%, 2,5% έτσι. Πρέπει να το δούμε βέβαια ακόμα. Αλλά αυτή είναι η εκτίμηση. Επίσης, Είπατε ότι ο κόσμος, οι πολίτες πρέπει να νιώσουν τα ωφέλη από το ευρώ. Έχετε δίκιο. Και αν τα σχόλιά μου φάνηκαν κάπως αρνητικά για κάποιους, λάθος. Λυπάμαι. Στη Νομισματική Ένωση όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να τηρούμε τα συμφωνημένα, προκειμένου να λειτουργήσει. Άρα η αλληλεγγύη συνοδεύεται από κανόνες. Αυτό ήθελα να πω, αυτό είναι που λέω πάντα και είναι σημαντικό. Τα πρώτα χρόνια του ευρώ ήταν πολύ καλά για όλους μας. Είναι αλήθεια, οι οικονομίες μας άνθησαν τα πρώτα 7 χρόνια και μετά περάσαμε στην επόμενη κακή επταετία, ελπίζω όχι άλλο, σε ένα δύσκολο οικονομικό κλίμα. Τώρα πιστεύω ότι αρχίζει να βελτιώνεται πια η κατάσταση. Κάποιος με ρώτησε, δεν είμαι σίγουρος, ο κύριος Κουντής ήτανε, για τις προτάσεις όσον αφορά τη συνταξιοδότηση, αν έρχονται από την ελληνική κυβέρνηση οι μεταρρυθμίσεις ταξιδιωτικές έγιναν σε συνεργασία με τους θεσμούς. Το καλοκαίρι του 2015 ήταν ένα στοιχείο κλειδί πάνω στο οποίο διαπραγματευτήκαμε το πρόγραμμα συμμετείχα σε κάποιες από αυτές τις συζητήσεις. Ε, πρόκειται για διαπραγματεύσεις, πραγματικά διαπραγματεύσεις μεταξύ των διαφόρων πλευρών. Δεν ήταν κάτι που επιβλήθηκε από τη μία πλευρά. Όχι. Έγιναν διαπραγματεύσεις προκειμένου να γίνει βιώσιμο το συνταξιοδοτικό και με τρόπο που να είναι αποδεκτός και από τους Έλληνες. Αναφερθήκατε και στο κούρεμα στην Κύπρο και πώς το βλέπω. Και η επόμενη ερώτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Λέτε κατά πόσο συμφωνώ με τον Όλυ Ρεν που είπε ότι το πρώτο πρόγραμμα έγινε για να στηριχθούν οι τράπεζες. Κοιτάξτε, στο πρώτο στάδιο της κρίσης στις χώρες μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ε, βέβαια η τράπεζα. Είχαμε τραπεζική κρίση, δημοσιονομική κρίση και χρησιμοποίησαμε πολλά από τα χρήματα του φορολογούμενου, με λάθο τρόπο κατά τη γνώμη μου, για να σώσουμε τις τράπεζες. Και ο κόσμος που επέκρινε τα πρώτα χρόνια του ελληνικού προγράμματος λέγοντας ότι μα όλα έγιναν μόνο για τις τράπεζες, έχουν κάποιο δίκιο. Και αυτό ισχύει για όλε μας τις χώρες. Οι τράπεζες παντού στην Ευρώπη σώθηκαν σε βάρο του φορολογούμενου. Γι' αυτό και φτιάξαμε την Τραπεζική Ένωση τώρα με υψηλότερες προδιαγραφές, με καλύτερη εποπτεία, με ένα πλαίσιο εξυγίανσης, διάσωσης, αν οι τράπεζες έχουν απώλειες. Ακριβώς για να μην ξαναβρεθούμε σε αυτή την κατάσταση. Το υψηλό δημοσιονομικό χρέος χωρών, που παραμένει σε πολλές ε, περιπτώσεις, έχει να κάνει με την τραπεζική κρίση και αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Μετά, τι άλλο. Υπήρξαν και ερωτήσεις για την ομάδα εμπειρογνωμόνων και τις συμβουλές τους των σοφών. Έγιναν συστάσεις για 11 τομείς. Για κάποιους από αυτούς οι εμπειρογνώμονες δεν συμφωνούσαν, δεν κατέληξαν ομόφωνα. Για άλλους τομείς συμφώνησαν όλοι. Ένα θέμα, το έθιξα ήδη μετά από την παρέμβαση της κυρίας Γιονγκέριους, θα ακολουθήσουμε τη σύστασή του στο τέλος του προγράμματος. Υπάρχει ένα συμβιβασμός δηλαδή ανάμεσα στους αρχικούς στόχους του προγράμματος και την ε, η υλοποίηση και το πώς θα προχωρήσουμε με τις συλλογικές συμβάσεις. Κάποιες άλλες συστάσεις τις επεξεργαζόμαστε τώρα, αποτελούν μέρος της τρίτης αξιολόγησης. Διάφορα μέτρα και μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη εφαρμοστεί ή αποτελούν μέρος της τρίτης αξιολόγησης. Οπότε έχουμε χρησιμοποιήσει καλά τις συστάσεις των σοφών. Ρωτήσατε κατά πόσο το Συμβούλιο Απασχόλησης πρέπει να εμπλέκεται ή όχι. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν να κάνουν ε, με ένα ευρύ πεδίο θεμάτων στις ε, κοινωνίες των χωρών που βρίσκονται σε πρόγραμμα. Πολλοί θεσμοί και η Επιτροπή και το ΑΕΜΕΦ βέβαια συμμετέχουν και έρχονται στο Eurogroup με ένα πακέτο συμφωνημένο μεταξύ των θεσμών και των λογοχωρών. Και πιστεύουμε ότι είναι αυτά τα οποία χρειάζονται για να ξαναμπεί στην κανονική ροή χώρα. Βάση τέτοιας συμφωνίας χρηματοδοτούμε στη συνέχεια τη χώρα μέσω του ESF πριν, του ESM τώρα. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Δεν προβλέπεται συμμετοχή κανένα άλλου συμβουλίου. Θα μπορούσε επί τη ουσία. Αλλά προ το παρόν ο σχεδιασμό του προγράμματος γίνεται ανάμεσα στου θεσμού και τη χώρα. Και μετά οι Υπουργοί Οικονομικών αποφασίζουν για τη χρηματοδότηση της χώρας που ζητάει ενίσχυση. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Για τον κύριο Βάλε. Είπατε πότε θα έχουμε τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις για τα μεγάλα ζητήματα. Αναφερθήκατε στις ανισορροπίες που έχουμε στην Ευρωζώνη. Εδώ θα έλεγα ότι οι ανισορροπίες αυτές στην Ευρωζώνη και μεταρρυθμίσεις χρειάζονται σε επίπεδο μακρό. Αλλά εξακολουθούμε όμως να χρειαζόμαστε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στις επιμέρους χώρες. Όχι μόνο στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα όχι μόνο σε, στις χώρες της Ευρωζώνης, σε όλες τις χώρες. Και αν θέλετε μάλιστα να διορθώσετε τις ανισορροπίες λογαριασμών, τρεχουσών ε, λογαριασμών με τα πλεονάσματα που υπάρχουν σε κάποιες χώρες, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και σε αυτές τις χώρες με πλεονάσματα. Χρειάζονται υψηλότερη μισθή σε αυτές τις χώρες. Στην Ολλανδία, στη Γερμανία για παράδειγμα, όπου οι μισθοί θα έπρεπε να αυξηθούν, θα βοηθούσε αυτό αλλά χρειάζονται και επενδύσεις. Σε υποδομές, στην εκπαίδευση, στην έρευνα. Θα βοηθούσε κάτι τέτοιο. Οπότε, ναι, χρειάζεται περισσότερη δουλειά επιμέρους, ναι, γίνεται η συζήτηση αυτή στο Eurogroup και ναι, όλο και περισσότερο τα πέντε χρόνια που είμαι στο Eurogroup, ναι, επιμείναμε πάρα πολύ στα δημοσιονομικά προβλήματα, αλλά όλο και περισσότερο τώρα στρεφόμαστε στις μεταρρυθμίσεις της Ευρωζώνης γενικότερα. Συζητάμε όλο και περισσότερο για την Τραπεζική Ένωση που είναι μέρος της μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης. Μιλάμε για το EDIS που είναι και αυτός ένας τρόπος να υπάρξει εξισορρόπηση στις διαφορές μεταξύ των χωρών μελών μας. Οπότε αυτού του είδους οι μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης ναι, πρέπει να συνεχιστούν όχι όμως αντί για τις εθνικές μεταρρυθμίσεις, αλλά ως συμπλήρωμα στις εθνικές μεταρρυθμίσεις. Μίλησα για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για τις συλλογικές συμβάσεις. Τι άλλο. Εκφράσατε μια ανησυχία, δεν έγραψα το όνομά σας, συγγνώμη. Αναφερθήκατε στην ποιότητα των θέσεων απασχόληση. Είπατε ότι στην Ελλάδα είναι μόνο χαμηλών δεξιοτήτων. Δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν βλέπω γιατί. Το βασικό για την Ελλάδα σήμερα είναι η ανάκτηση εμπιστοσύνη στη χώρα, στην οικονομία, αλλά και στο διοικητικό πλαίσιο, στο νομικό σύστημα, έτσι ώστε όλο και περισσότερες επενδύσεις να επιστρέψουν στη χώρα. Και σίγουρα αν γίνουν οι επενδύσεις, τότε αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται και καλύτερες δεξιότητες, πιο σύγχρονες, αυτές που χρειάζονται στο σημερινό κόσμο. Οπότε και για την ποιότητα της απασχόλησης και για την ποσότητα της απασχόλησης χρειάζονται επενδύσεις. Αρχίζει να γίνεται αυτό. Βλέπουμε ότι αρχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον απ' έξω, αλλά το κλειδί σε όλα αυτά είναι η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα. Αναφέρθηκα επίσης στις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη και τέλος, κύριε Παπαδημούλη, όντω συζητάμε πολύ συχνά για την Ελλάδα και όπως πολύ σωστά είπατε, συχνά διαφωνούμε μεταξύ μας. Αλλά εδώ νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε για το ότι η προοπτική είναι πολύ καλύτερη σήμερα από ό,τι κατά το παρελθόν. Και αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επικοδομητικά όπως κάνουμε τώρα, πράγματι αυτό θα δείξει ότι κάτι αλλάζει και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας. Η τρίτη αξιολόγηση, από ό,τι μου λένε ακόμα και σήμερα, οι θεσμοί πάνε καλά τα πράγματα. Σίγουρα χρειάστηκε, μάλλον χρειάζονται ακόμα πολλά, να εφαρμοστούν πολλά, αλλά γίνονται πολλά στην Ελλάδα και έχει δεσμευτεί υπέρ αυτών η ελληνική κυβέρνηση, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να δώσουμε ξανά χρήματα στην Ελλάδα, να εκταμιεύσουμε δηλαδή, στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Και για τη συζήτηση όσον αφορά το χρέο, θα θυμόσαστε ότι η τελευταία μα συμφωνία ήταν να υπάρξει ένα μηχανισμό ο οποίο θα συνδέει ε, μέτρα ανακούφιση που εξαρτώνται από τι εκτιμήσει ανάπτυξη και τι επιδόσει τη Ελλάδα. Αν λοιπόν ε, και πάλι υπάρξουν κάποια σοκ ή υπάρξει χαμηλότερη επίδοση, ε, πάλι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μέτρα να ανακουφίσουμε ε, την Ελλάδα. Αυτός ο μηχανισμός θα είναι πάρα πολύ σημαντικός για την επόμενη δεκαετία και θα τον δούμε από την αρχή της επόμενης χρονιάς. Ε, σκέφτομαι πολύ θετικά ότι προχωράμε προς την λήξη του προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάσιλπλουμ. Περιμέναμε πολύ καιρό στην Επιτροπή μας ε, τη συνάντηση αυτή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ λοιπόν που ήρθατε εδώ. Είμαστε η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι λοιπόν σημαντικό να σας έχουμε στην ημερήσια διάταξή μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε και που προσπαθήσατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας και ελπίζουμε να επανέλθετε πριν τις ευρωεκλογέ και να μας δώσετε περισσότερα αποτελέσματα. Και ε, ακούτε τις δικές μας ε, ε, επικριτικές ερωτήσεις, αλλά και εμείς πάντα ακούμε τα καλά σας αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Επόμενη συνεδρία 21 Νοεμβρίου. 9 με 12.30. Συντονιστές έχουμε επίσης την ίδια μέρα. Σας ευχαριστώ για αυτήν την μακρά και επικοδομητική συνεδρίαση της Επιτροπής. Ευχαριστώ.